can we Αγαπητοί συναδελφοί, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε όλοι. Να καλωσορίσουμε και τους προσκεκλημένους μας που είναι έτοιμοι για να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ρόλο των δημοσίων βιβλιοθηκών. Πριν ε, συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω δύο λόγια ε, εισαγωγικά. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Αν δεν με ακούτε, μπορείτε να φορέσετε τα ακουστικά σας. Καταρχάς, γνωρίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι είναι καθοδόν, αλλά δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο, γιατί νομίζω ότι εκφράζω την άποψη όλων σας νιώθαμε ιδιαίτερο πόνο αυτή την εβδομάδα με την τραγική απώλεια, με τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας, μιας ε, νεαρής ε, Βρετανής ε, βουλευτού, της Τζο Κόξ, η οποία δολοφονήθηκε βάνασα στο Λονδίνο, ενώ ασκούσε τα καθήκοντά της στην εκλογική της περιφέρεια. Μια νέα γυναίκα η οποία νομίζω μας συγκίνησε όλους, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός, διότι προέχει ο άνθρωπος ο πόνος της οικογένειάς της, μια νεαρή οικογένεια με δύο παιδιά. Ε, η ίδια την Τετάρτη θα γινόταν 42 ετών και μια γυναίκα η οποία είχε ξεκινήσει από τον εθελοντισμό, εργαζόταν στην Oxfam, ήταν ε, υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσφύγων, ε, της ιδέας μιας αλληλέγγυας Ευρώπης ε, υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και φυσικά ένας άνθρωπος που είχε πολύ ε, ακέραιες αξίες και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε όλοι σε αυτό το στάδιο της δύσκολης ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα απλώ λοιπόν να πω ότι θεωρώ ότι πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτή τη γυναίκα, διότι είναι μια γυναίκα η οποία πλήρωσε ακριβό τίμημα την ίδια της τη ζωή, γιατί έλεγε ελεύθερα την άποψή της και ασκούσε ένα ευγενέ επάγγελμα ε, του πολιτικού τη ε, της βουλευτού. Ε, θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού υγιής μνήμη της. Grazie. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να περάσω στην έκρηση της ημερήσιας διάταξης. Απευθύνομαι στους συναδέλφους, αν δεν υπάρχουν στάσεις, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο και να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης Τη 18 και 19 Απριλίου, τα έχετε στα εγγραφά σας. Υπήρχε ένα τεχνικό λάθος ε, στα πρακτικά τις 18 και 19 Απριλίου. Πρέπει να γίνει μια προστίκη, θα διορθωθούν τα πρακτικά και θα τα εγκρίνουμε στα συνεδρίες του Ιουλίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ε, για αυτά τα πρακτικά για τις 25 και 26 Απριλίου, ε, μπορούμε να εγκρίνουμε τουλάχιστον αυτά. Υπάρχει διερμηνία σήμερα σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, τα οποία μπορείτε και να μιλήσετε και να ακούσετε. Η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται ζωντανά μέσω web streaming ε, στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και στις αποφάσεις ε, των συντονιστών που ελήφθησαν στις 20 Μαΐου. Τις μάθατε, σας εστάλησαν ε, τα πρακτικά ε, στις 30 Μαΐου και εγκρίνονται γιατί δεν υπήρξε καμία ένσταση από καμία πολιτική ομάδα. Να φτάσουμε τώρα στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ακρόαση που ζήτησαν αρκετοί από εσά, διότι θεωρούμε ότι το να αναφερόμαστε σήμερα στην πρόσβαση στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά δικαιώματα, να αναφερθούμε και σε αυτά, στον αλφαβητισμό, καθώς επίσης και στο νέο ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο των ε, δημοσίων βιβλιοθηκών, το οποίο ε, κάνει πολύ σημαντικές δράσεις ε, και εκστρατείες προώθησης, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς ως Ευρωβουλευτές και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να σταθούμε και να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Φρονώ ότι σήμερα αλλάζουν ε, τα πράγματα και λόγω ψηφιακή εξέλιξη, αλλά και για αυτό το οποίο αντιπροσωπεύουν ως ε, πολιτιστικά αγαθά, τα οποία βοηθούν και στην κοινωνική ένταξη. Θα θέλαμε να κατανοήσουμε λοιπόν πού ε, τοποθετούνται σήμερα οι δημόσιες βιβλιοθήκες, πώς έχει αλλάξει ο ρόλος τους, ποιες είναι οι προκλήσεις και αυτό φυσικά θα γίνει με παρουσία κάποιων εμπειρογνωμόνων, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την σημερινή τους παρουσία. Εδώ εξ αριστερών μου λοιπόν έχουμε την κυρία Μπάρμπαρα Λίζον, που είναι η Διευθύντρια της ε, ε, Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Μπρέμα. Συμμετείχε και στα ε, δημόσια θέματα της ε, οργάνωσης των επαγγελματικών βιβλιοθηκών και φυσικά θα μας δείξει πώς ε, οι δημόσιες βιβλιοθήκες σήμερα αποτελούν τμήμα του πολιτιστικού ε, τοπίου του 21ου αιώνα και μπορούν να διαδραματίσουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο δεύτερος εμπρογνώμονο είναι ο Φρανκ Βίσμαν από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ο οποίος θα μας πει πώς οι βιβλιοθήκες θα εμβαθύνουν και πώ συνεισφέρουν στην εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνία, επομένω θα αναφερθούμε περισσότερο στις δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται σήμερα, προκειμένου να υπάρχει και η δυνατότητα να ερμηνεύσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες προσφέρονται αφιδώς. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Dan Mount, ο οποίος έχει ε, συντάξει αρκετά σημαντικές εκθέσεις που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό δανεισμό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα του ηλεκτρονικού δανεισμού, του e-lending και θα μας εξηγήσει διάφορες σημαντικές ε, μεθόδους ε, δανεισμού και μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων και μέσα από διάφορες πλατφόρμες και μας εξηγούν πώς οι διάφορες ε, δημόσιες βιβλιοθήκες διαθέτουν τις διάφορες δημοσιεύσεις τους και τα βιβλία που έχουν και στην Ευρώπη αλλά και στην Βόρεια Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα οποία θα μας πούν οι εμπειρογνωμονές μας και τους ευχαριστώ πολύ. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην κυρία Λίζου για να παρέμβει στη συζήτησή μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για το ρόλο των δημοτικών βιβλιοθηκών στις τοπικές κοινωνίες των 21 ου αιώνα. Πρέπει να συνηθίσω αυτό το πρόγραμμα εδώ. Βλέπετε τη δομή της παρουσίασής μου εν μέρει αφορά όχι μόνο τη δομή, αλλά και θα ακούσετε κάποιες δηλώσεις. Κάποιες δηλώσεις ε, που αφορούν γιατί ε, είναι τόσο σημαντικές οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι δημοτικές βιβλιοθήκες και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση τους. Ας αρχίσουμε όμως με το τι συμβαίνει στο ε, παρασκήνιο. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες ανήκουν στις τοπικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν ε, αρμοδιότητα αυτών των τοπικών αρχών και αυτό ε, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο λόγω των ανισοτήτων παρατηρούνται σε μια κοινότητα. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες τους να λαμβάνονται υπόψη και ως προς τις ανισότητες. Υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που συντελούνται και ε, όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και όσον αφορά την ε, νέα κοινωνία που εμφανίζεται. Και πρέπει λοιπόν οι πολίτες να προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα κοινωνία και η κοινωνία σε αυτούς. Ορισμένοι συνάδελφοι έκαναν μία σύγκριση και ε, θεώρησαν ότι η, επινοή, η, η εφεύρεση της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει τώρα με την ψηφιακή επανάσταση. Χρειάζεται λοιπόν νέα πολιτική, αποτελεσματική πολιτική για την εκπαίδευση και πρέπει να καταλάβουμε ε, ποια εργαλεία είναι χρήσιμα για αυτές τις εξελίξεις. Ας δούμε τώρα τις δημοτικές βιβλιοθήκες και πώς αυτή ε, η κατάσταση φαίνεται σε αυτές. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι εύκολα κατανοητές από τους πολιτικούς. Ε, ορισμένοι συνάδελφοι πολύ συχνά με ρωτούν γιατί οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι τόσο σημαντικές, αφού υπάρχει το διαδίκτυο. Και ε, επίσης υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί των ε, τοπικών αρχών, υπάρχουν περικοπές στο δημόσιο και επειδή οι δημόσιες υπηρε... Ε, βιβλιοθήκες είναι κατά κύριο λόγο θελοντικές, οι περικοπές τις πλήττουν. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει μείωση ε, των βιβλίων που δανείζονται, όμως αυτό ανήκει στις στατιστικές που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Φυσικά υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από τους πολίτες για ψηφιακές υπηρεσίες, γι' αυτό οι βιβλιοθήκες πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, όπου ε, θα τις καθιστούν ελκυστικές για τους πελάτες τους, για τους χρήστες. Ας αρχίσουμε όμως ε, με το ρόλο της δημόσιας βιβλιοθήκης ως σημαντική πύλη προς την κοινωνική συμπερίληψη, την κοινωνική ένταξη. Οι δημόσιε βιβλιοθήκε πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των πολιτών και να στηρίζουν τη γνώση μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν. Ακριβώς διότι υπάρχει η δυνατότητα σε αντιδιαστολή με τα σχολεία μια δημόσια βιβλιοθήκη να ε, χρησιμοποιείται από το άτομο για όλη του τη ζωή οι καλές δημόσιες βιβλιοθήκες ε, πολλές φορές θεωρούνται τρίτο σπίτι, μετά το σχολείο, μετά τη δουλειά, μετά το σπίτι και πολλές φορές μάλιστα ε, αναφέρονται στη Συγκαπούρη συγκεκριμένα ως ε, δεύτερο σαλόνι. Οι βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος λοιπόν όπου αισθάνεται κάποιος ευχάριστα και φυσικά ευνοούν την μη τυπική και άτυπη μάθηση. Εδώ βλέπετε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε το project Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2020. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν περίπου 100 εκατομμύρια επισκέπτες και όχι ε, και αυτοί δεν είναι όλοι, είναι μόνο όσοι έχουν αιτήσια κάρτα μέλους. Ο πραγματικό αριθμό είναι μεγαλύτερος δηλαδή. Βλέπουμε εδώ και κάποια στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν ε, το πώς επηρεάζουν οι βιβλιοθήκες τις πιθανότητε έβρεση εργασία από τους πολίτες όταν εκείνοι ψάχνουν δουλειά ή προσπαθούν να επεκτείνουν τις ε, γνώσεις τους. Βλέπουμε λοιπόν πολύ εντυπωσιακά νούμερα. Βλέπουμε εδώ ότι τα αποτελέσματα της ε, βιβλιοθήκης στη δημιουργία δεξιοτήτων και ε, επαγγελματικών προσόντων. Εδώ να σας ε, αναφέρω κάποια επιχειρήματα που στηρίζουν τις διαφάνειες. Εδώ αυτές οι φωτογραφίες ε, μας δείχνουν τους διαφορετικούς ρόλους που παίζει μια ε, δανειστική βιβλιοθήκη. Βλέπουμε πώς μπορεί να βοηθήσει διάφορες ομάδες ανθρώπων, ε, μετανάστες, βλέπουμε κάποιοι που κοιμούνται εκεί, βλέπουμε νέους που διαβάζουν ε, ή βλέπουν ψηφιακά ψηφιακό περιεχόμενο. Ο κύριος βέβαια πυρήνας είναι τα βιβλία. Τώρα, οι δημόσιες βιβλιοθήκες τώρα παρέχουν μια ευρύτατη γκάμα υπηρεσιών. Δεν δανείζουν μόνο βιβλία, αλλά έχουν κατανοήσει το γεγονό ότι πέρα από το δανεισμό βιβλίων και άλλων ε, οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να προσφέρουν μια πληθώρα υπηρεσιών για να εξυπηρετήσουν τι ε, ανάγκε του κοινού. Ανάλογα βέβαια με τις εξελίξεις μιας ε, κοινότητας και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Νομίζω πως μου λείπουν κάποιες διαφάνειες εδώ. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εικόνες για να δείτε και στην πράξη. Θα βλέπατε λοιπόν, αν είχα αυτές τις ε, διαφάνειες, ομάδες παιδιών που διαβάζουν σε iPad, υποβοηθούμενα από βιβλιοθηκάριους. Α, ε, μου λείπει και άλλη εικόνα βλέπω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Οι βιβλιοθήκες όμως είναι πολύ σημαντικές στην ενσωμάτωση και συμπερίληψη του κοινού βλέπουμε ότι είναι μία υπηρεσία άμεσης πρόσβασης, είναι πολύ εύκολο να μπει σε μία δημόσια βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή να πάρεις κάποια πρώτερη έγκριση, εκτός από το να έχεις μαζί σου την κάρτα της βιβλιοθήκης. Μπορείς λοιπόν με αυτή την κάρτα να έχεις αμέσω πρόσβαση στις υπηρεσίες. Τώρα, είναι δωρεάν η επίσκεψη. Ε, πολλές φορές η κάρτα κοστίζει, όμως πολλές φορές το κόστος ε, είναι μειωμένο ή τα παιδιά μπαίνουν ε, και μπορούν να δενίζονται βιβλία δωρεάν. Υπάρχει λοιπόν ε, άμεση πρόσβαση με μηδαμινό ή ελάχιστο κόστος για το κοινό. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι νέο. Οι βιβλιοθήκες ανέκαθεν προσπαθούσαν να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση όλων των πολιτών σε μια κοινωνία. Θυμηθείτε ότι τη δεκαετία του 50 όταν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι έφεραν τις δημόσιες βιβλιοθήκες στην βιβλία στη Γερμανία Γερμανία, οι βιβλιοθήκες είχαν αυτόν τον σκοπό, την ενσωμάτωση, την ένταξη, τον εκδημοκρατισμό ε, του κοινού. Τώρα, η πρόκληση που έχουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες που έχουν έρθει σε μεγάλους αριθμούς στην Ευρώπη. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς γιατί είναι μια υπηρεσία άμεσης πρόσβασης και ανέλαβαν αυτό το ρόλο και έχουν ήδη αναπτύξει νέες υπηρεσίες οι οποίες ε, ολόνα και αναπτύσσονται για τους πρόσφυγες. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες της βιβλιοθήκης μου στη Βρέμη. Βλέπετε άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν που βρίσκονται ε, σε διάφορους χώρους μάθησης. Βλέπετε εδώ μια βιβλιοθηκάριο που μιλά με μετανάστες, πρόσφυγες και τους δείχνει συγκεκριμένα βιβλία που βοηθούν στην εκμάθηση της νέας τους γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στη γερμανική κοινωνία. Σε πολλές βιβλιοθήκες υπάρχουν υπολογιστές όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει πάνω από 2.000 ημερήσιες βιβλιοθήκες. Όταν λοιπόν φτάνει σε μια ξένη χώρα έχεις πρόσβαση ε, στον τύπο. Και είναι ένας χώρος ε, επίσης που μπορούν να φιλοξενηθούν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, εκτός από τους παραδοσιακούς χώρους φιλοξενίας. Τώρα υπάρχουν και άλλες διαστάσεις σε μια βιβλιοθήκη. Πολλοί ε, θεωρούν πως ε, το κόστος είναι υψηλό και πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κόστους ε, σε μια δημόσια βιβλιοθήκη. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση της βιβλιοθήκης του Τορόντο, προσπάθησαν να δουν τις άμεσες δαπάνες μιας της βιβλιοθήκης και τα άμεσα και έμεσα ωφέλη αυτής. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μόνο. Μπορείς ε, εδώ λοιπόν να εισαγάγεις τα χρήματα που δαπανούνται και να δεις το αποτέλεσμα. Φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ ε, επιφανειακό προς το παρόν, όμως βλέπουμε ότι για κάθε δολάριο Καναδά που επενδύθηκε το, το όφελος ήταν 6 δολάρια Καναδά. Αυτό βλέπουμε να έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείες, στη Φλόριδα συγκεκριμένα. Και φυσικά προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, όμως ε, εδώ βλέπουμε ότι για κάθε δολάριο ή ευρώ που επενδύεται, το, ε, η απόδοση, το όφελος είναι πολύ υψηλότερο. Ας περάσουμε όμως τώρα στα αποτελέσματα, στα βασικά αποτελέσματα μιας δημόσιας βιβλιοθήκης. Δημιουργούν υποδομές για, για τον πολιτισμό, τη μάθηση, τη γνώση και την εκπαίδευση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα καθιερωμένο ε, ίδρυμα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να χτίσεις από το μηδέν. Και πολλές φορές ε, περιμένουμε από τους ε, πολιτικούς να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες υποδομές. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι βιβλιοθήκες είναι μεγάλος ε, παράγοντας στην ε, δημιουργία συνεργασίας. Χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες για να διευκολυνθεί η συνεργασία ανάμεσα σε άλλα ιδρύματα, σε άλλους οργανισμούς. Στη Βρέμη, για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη μας συνεργάζεται με το 100% των σχολείων του κρατηδίου. Και αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που έχει άμεσο όφελος. Τώρα, θα ήθελα να σας δείξω και το εξής. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει μία ε, επανεξέταση του ρόλου της δημόσιας βιβλιοθήκης. Εδώ βλέπετε όλες τις ε, κατηγορίες που ε, συζητούνται στις κατοχώρες, για παράδειγμα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι οι βιβλιοθήκες έχουν το δυναμικό για να γίνουν στο μέλλον ηγετική ε, φυσιγνωμία σε μια κοινότητα. Τώρα, όσον αφορά την Ήπεθρο και τις ε, μικρές πόλεις, ε, γνωρίζετε ότι λόγω της ανεργίας, λόγω της έλλειψης πολιτιστικών δραστηριοτήτων πολλοί εγκαταλείπουν αυτά τα μέρη και πολλές φορές η βιβλιοθήκη είναι ο μόνος χώρος πολιτισμού σε ένα μικρό μέρος, σε ένα χωριό, μια πόλη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές οι κινητές μονάδες είναι μια λύση. Εδώ ένα παράδειγμα από τη Ρουμανία. Υπάρχει ένα project, το Biblionet Apia, το οποίο στηρίζεται από το Ίδρυμα Gates και είναι ένα παράδειγμα του πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να ε, επιτύχουν τους ε, βασικούς στόχους πολιτικής. Πώς μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν τους αγρότες να πουλήσουν τα προϊόντα τους ε, με καλύτερη τιμή. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το περίμενε κανείς, όμως όντως συνέβη λόγω της βιβλιοθήκης. Επίσης, οι βιβλιοθήκες είναι κεντρικά σημεία αναφοράς σε μία πόλη σε ένα μέρος όσοι χρησιμοποιούν μια βιβλιοθήκη φέρνουν κίνηση. Για παράδειγμα, στη Γερμανία 180 εκατομμύρια επισκέπτες ε, το χρόνο ε, πηγαίνουν σε μια δημόσια βιβλιοθήκη είναι περισσότεροι από όσους πηγαίνουν στα γήπεδα σε αγώνες πρώτης εθνικής. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Επίσης, ε, ανάπτυξη αστική Είναι το τελευταίο μέρος της παρουσίασής μου και θα ήθελα εδώ να σας δείξω ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Είναι το κατάστημα Idea στο Λονδίνο, το οποίο βρίσκεται σε ένα μέρος το οποίο δεν ε, είναι σε καλή περιοχή και είναι μια βιβλιοθήκη. Ερωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι πώς θέλετε να είναι αυτή η βιβλιοθήκη, η οποία στη συνέχεια δημιουργήθηκε με βάση τις ε, προτάσεις του κοινού. Και αυτή η βιβλιοθήκη έχει προσελκύσει κόσμο στο μέρος αυτό. Στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, είχαμε μια παρόμοια περίπτωση. Χτίστηκε μια βιβλιοθήκη πάνω στις παλιές γραμμές του τρένου. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κεντρική βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη που θα είναι υπόδειγμα και θα μπορούν να βασίζονται σε αυτή και άλλες μικρότερες. Τώρα, ε, τη βιβλιοθήκη που σας έδειξα στην εικόνα την έχει χτίσει ένας από τους πιο διάσημους αρχιτέκτονες αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Άρχου στη Δανία που άνοιξε το 2015. Ε, χτίστηκε πάνω σε παλιές λιμενικές εγκαταστάσεις και εδώ θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα είδος σύνδεσης ανάμεσα στο, στην πόλη και στο λιμάνι. Και καταλήξαμε στη βιβλιοθήκη του Άρχους. Η τελευταία μου, πρώτη τελευταία μου διαφάνεια ε, περιλαμβάνει κάποιες προτάσεις. Ελπίζω να μπόρεσα να σας δείξω την σημασία που έχει μια βιβλιοθήκη και για την κοινωνία και για το άτομο. Η δουλειά μας όμως θα μπορούσε να πάει πέρα από αυτό και να γίνει πιο αποτελεσματική εάν είχαμε και την πολιτική στήριξη. Γι' αυτό ελπίζω οι προτάσεις και οι συστάσεις αυτές να έχουν τη στήριξη στην νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως ε, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια νομοθεσία που να προωθεί γενικότερες ιδέες για τις βιβλιοθήκες. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Πέρα από τη δουλειά σας, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μεταγισματισμός του ρόλου των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη. Και μου αυτή η ιδέα σας ε, ότι λειτουργούν υποστηρικτικά και προσελκύουν τους ε, χρήστες οι βιβλιοθήκες τόσο σε ε, αστικές όσο και περιοχές όσο και στην Ήπεθρο. Σίγουρα θα έχουμε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ο Φρανκ μας ακολουθεί τώρα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Άμστερνταμ για την προώθηση της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία στις δημόσιες βιβλιοθήκες. θα ήθελα να κάνω μια σύντομη επισκόπηση αυτή της ε, έννοια, της ε, πρόθεση παιδεία τα μέσα και της πληροφορίας ε, στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Θα ήθελα να μιλήσω για, αυτή, ε, για τον ορισμό αυτής της έννοιας, για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία και στη συνέχεια να περάσω σε αυτά που έχουν κάνει και θα κάνουν οι βιβλιοθήκες για την πρόθεση αυτής της παιδείας. Ε, κατόπιν θα σας παρουσιάσω κάποιες προσεγγίσεις ε, όπως έχουν υιοθετηθεί από διεθνούς οργανισμούς και Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών προσπαθειών που γίνονται για την παιδεία στα μέσα και τις πληροφορίες και θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Τι εστί λοιπόν παιδεία στα μέσα και την πληροφορία. Δεν έβαλα καθόλου φωτογραφίες, ευτυχώς κιόλας. Διαβάζω τον ορισμό. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, αλλά βασικά είναι η ικανότητα κάποιου να έχει μία διάδραση, ε, να έχει απαιτούμενε δεξιότητες για να έχει μία διάδραση με, τις, ε, με τα μέσα ενημέρωσης ε, και την πληροφορία. Είναι η κριτική εξολόγηση της πληροφορίας, αν θέλετε και βάση ε, σύνομων και ηθικών προτύπων. Στη συνέχεια, όταν μιλάμε για την παιδεία στην πληροφορία, ε, είναι από ιστορικής πλευράς επίσης πολύ διαφορετική έννοια. Πρώτον, αναγνωρίζετε εσείς ο ίδιος πότε χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να δράσετε στην καθημερινή σας ζωή. Και αυτή τη στιγμή εντοπίζετε αυτή την ανάγκη σας, πρέπει να εντοπίσετε και τις προφορές, να τις αξιολογήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για την εξυπηρέτηση των ε, δικών σας ε, στόχων. Ε, είναι πολύ διαφορετική η ιστορική πορεία αυτών των δύο ενιών. Η παιδεία στα μέσα έρχεται από τους εκπαιδευτές, ενώ η παιδεία της πληροφορίας ε, προέρχεται από αυτό το πεδίο των δημοσίων βιβλιοθηκών. Βλέπουμε όμως μια συγχώνευση αυτών των ενιών τη σήμερα ημέρα και μπορεί να αποδοθεί αυτό στο ότι έχουν συγχωνευτεί και οι δομές των μέσων και της πληροφορίας ε, στο ψηφιακό περιβάλλον. Η ψηφιοποίηση των πληροφοριών έχει οδηγήσει οδηγεί σε προσέγγιση της παιδείας πληροφορίας και της παιδείας στα μέσα. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες από το, τη δεκαετία του 70 στον περασμένο αιώνα ε, ε, προωθούν την παιδεία και ε, βοηθούν τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές να εντοπίζουν και να αξιολογήσουν πηγές πληροφοριών. Ε, θα μου πείτε, μα τα ξέρουν όλα οι δάσκαλοι. Μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει και μπορεί να μην έχουν οι ίδιοι ανάγκη για κάποιες πληροφορίες, αλλά ε, αναγνωρίζουν την αξία ενός βιβλιοθηκάριου παραδείγματο χάρη όταν ε, αναζητούν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Ε, τώρα, σε σχέση με τις σχολικές ε, βιβλιοθήκες. Γενικά μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναφερθούμε και στην συμβολή των σχολικών βιβλιοθηκών στο κίνημα αυτό. Ε, στα προς τα τέλη του περασμένου αιώνα υπήρξε η προώθηση των δεξιοτήτων ε, στις τεχνολογίες των πληροφοριών μέσα από τις δημοσίες βιβλιοθήκες ε, για τα παιδιά και για τους ενήλικες ε, και όλοι επωφελήθηκαν από τέτοια προγράμματα. Για την παιδεία στα μέσα και την όλη συζήτηση υπάρχουν ε, δύο ε, προσεγγίσεις, να το πούμε έτσι. Κάποιοι το εξετάζουν από τη σκοπιά της προστασίας, αυτό κυρίως όταν μιλάμε για το δημόσιο διάλογο και την εκπόνηση πολιτικής, ε, πώς μπορείτε δηλαδή από τα ε, ιονή αρνητικά αποτελέσματα των μέσων της πληροφορίας να προστατεύσετε τους πολίτες και στον αντίποδα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αξιοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που βρίσκονται εκεί για ε, τους δικούς σας ε, σκοπούς. Στο δεύτερο τμήμα εντοπίζεται ο ρόλος περισσότερο των ε, δημοσίων βιβλιοθηκών διότι ε, κάποιος που έχει την δυνατότητα και τις δεξιότητες μπορεί να έχει μια υγιή ε, διάδραση και να ε, λειτουργεί αυτόνομα και να προστατεύει τον εαυτό του όταν χειρίζεται αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, οι βιβλιοθήκες δεν είναι μόνο σημεία πρόσβασης ε, στις πληροφορίες, αλλά ολοένα και περισσότερο με εξελίσσονται σε κέντρα ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Δεν ε, είναι μόνο ο υπάλληλο βιβλιοθήκη που σα βοηθάει να βρείτε, να εντοπίσετε τι πληροφορίε, ε, αλλά λειτουργεί και ω σημείο σύνδεση για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Μαθαίνουν εξάλλου και αυτοί οι άνθρωποι από τα μέλη τη κοινότητα. Και αυτό τους βοηθά και στην καθημερινή τους δουλειά, ε, όταν ε, παραδίνουν μαθήματα, παραδείγματο χάρη, για την παιδεία για ε, τους υπολογιστές. εργαστήρια μέσων, επιμορφωτικά εργαστήρια, παραδείγματο χάρη, media labs, πώς χρησιμοποιεί κάποιος το iPad, το iPhone, χρήση λογισμικών, ε, βοήθεια για να μπορέσει να μάθει κάποιος πώς μπορεί να φτιάξει ένα βίντεο και να το ανεβάσει στο YouTube και στο Vimeo. Ε, δεν μαθαίνει κάποιος μόνο διαβάζοντας αλλά και ε, κάνοντας, περνώντας στη, στην πράξη και με αυτά τα maker spaces, ε, ε, τους ε, χώρους δράσης των βιβλιοθηκών, με τη χρήση αυτών των νέων gadgets, με τη χρήση των νέων υπολογιστών και των νέων συσκευών, βοηθούν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που έχουν και πλάκα, αλλά πέραν αυτού βοηθούν για να μπορείτε ε, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για την καθημερινή σας ζωή. Έχουμε και τα περίφημα ε, hackathons, ε, σχεδιαστές υπολογιστών και χρήστες έρχονται σε επαφή για να δημιουργήσουν νέα πράγματα, να φτιάξουν νέους καταλόγους εμπλουτισμένους από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο για τις ίδιες τις βιβλιοθήκες, παραδείγματος χάρη. Ε, αυτό είναι το δυνατό σημείο των βιβλιοθηκών, λοιπόν, παιδεία σε πληροφορίε. Ε, ε, οι ερευνητέ τώρα στον ακαδημαϊκό κόσμο προσπαθούν να τυποποιήσουν, ε, αν θέλετε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για να υπάρχουν οι ορισμοί τη της παιδείας στην πληροφορία, στα μέσα και... Αυτή η έννοια της παιδείας στην πληροφορία χρησιμοποιείται πλέον και από πολλές, ε, πολλά κράτη-μέλη, πολλές κυβερνήσεις για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνεται πλέον αυτή ε, η έννοια στα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Επιτροπή και ο ΣΑ έχουν προωθήσει κυρίως ε, τις ψηφιακές δεξιότητες. Βέβαια δεν είναι το ίδιο αυτό με την παιδεία στην πληροφορία, αλλά ε, και το εξετάζουν από μια διαφορετική σκοπιά. Όμως η, η Διεθνής Ένωση των ε, Βιβλιοθηκών και η UNESCO παραδείγματος χάρη έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν αυτή την έννοια να προσδώσουν μάλλον μια νέα πολιτιστική εκπαιδευτική διάσταση σε αυτήν την έννοια. Και το 2012 κατέληξαν ε, και στην ε, δήλωση της ε, Μόσχας και παραθέτω, γιατί ξανά είπαμε ότι είναι ολιστική έννοια παιδεία στα μέσα και τις πληροφορίες, γνώσεις, στάσεων, πρακτικές, και ούτω καθεξής που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παραγωγή περιεχομένου με σύνομο τρόπο, με δεντολογικό τρόπο Νομίζω ότι είναι καλός αυτός ο ορισμός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την ε, προσέγγιση αυτών των ενιών παιδείας στα μέσα και της ε, πληροφορίας. Τι γίνεται τώρα με τα ε, εκπαιδευτικά προγράμματα. Λοιπόν, για την παιδεία την ε, πληροφορία. Δεν έχουμε παρακολουθήσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προγραμμάτων τόσο όσο έχουμε ερευνήσει την συμπεριφορά των χρηστών. Δηλαδή πώς στην καθημερινή του ζωή χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες ε, οι χρήστες ε, και αυτό είναι και σημαντικό για να είναι γράμματος κάποιος ε, στα, στην πληροφορία για τα παιδεία στα μέσα. Θα έλεγα ότι ακόμη δεν έχει κατοχυρωθεί αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και αυτό μπορεί να αποδοθεί στις πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, θεωρητικές ή πρακτικές, παραδείγματος χάρη. Παρόλα αυτά, Εν γέννη, αποτιμώντα αποτελεσματικά τα προγράμματα, δεν είναι βεβαίω οι δημόσιε βιβλιοθήκε ε, τόσο γνωστέ ε, οι πληροφορίε και όχι επειδή δεν έχει παρακολουθηθεί ε, και αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, αλλά έχει γίνει αυτό σε τοπικό επίπεδο και δεν έχουν ομογενοποιηθεί τα δεδομένα για να συνάξουμε συμπεράσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, όταν έχουμε ε, το πλαίσιο αξιολόγησης πάντως ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδυάζεται εκεί η θεωρία και η πράξη για τη συλλογή των δεδομένων, κατευθυντήριες γραμμές και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο οι βιβλιοθήκες αλλά και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί φορείς. Εάν γίνει αυτό θα μπορέσουμε με πιο σημαντικό τρόπο πλέον να συλλέγουμε τις πληροφορίες και να διαπιστώσουμε εάν ε, είναι ή όχι αποτελεσματικά τα προγράμματα και ε, ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνουμε, να, ε, ποιες βελτιώσεις πρέπει να επιφέρουμε στα προγράμματα για να τα καταστήσουμε αποτελεσματικότερα. Θα κατέληγα τώρα στο συμπέρασμα ότι αυτή η ομοιόμορφη προσέγγιση για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και αξίζει την υποστήριξή μας. Οι πολίτες από όλε τι ηλικίε ε, θα πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να έχουν τις ευετούμενε ε, δεξιότητες ε, για να προωθήσουμε την παιδεία τους στα μέσα και την πληροφορία για να προστατεύουν τους, ε, να αυτοπροστατεύονται από τις ενδεχομένως επιζήμιες ε, επιπτώσεις της χρήσης ε, των μέσων και της πληροφορίας και να γίνεται η χρήση των πληροφοριών με πιο διοντολογικό τρόπο. Θα έλεγα επίσης ότι είναι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη σημαντική συμβολή εδώ και χρόνια των δημοσίων βιβλιοθηκών ε, στον τομέα της παιδείας ε, στα μέσα και την πληροφορία. Πέραν αυτού, ε, σημαντική είναι η συμβολή των σχολείων και των γονέων. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και οι γονείς βοηθούν πολύ για την πρόθεση της παιδείας σε αυτούς τους τομείς και όσοι είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ενήλικες ε, μπορούν ε, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις και σε, αυτές, σε αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα για να αποκτήσουν τις δεξιότητες μέσα στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Λόγω περικοπών ε, σε πολλά κράτη-μέλη δεν υποστηρίζεται πολλές φορές αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστούν αυτά τα επιμορφωτικά εργαστήρια για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία. Ε, κατόπιν θα πρέπει να συνεχίσουμε με μια ενιαία προσέγγιση διότι πλέον έχουν, είναι μια ολιστική προσέγγιση αυτή που ακολουθούμε, δεν είναι πλέον δύο διακριτές έννοιες και έχουμε και τον ορίζοντα 2020 ε, στο οποίο μπορούμε να ε, χρησιμοποιώντας και το πλαίσιο της ε, UNESCO να συνεχίσουμε την προσπάθεια παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών για την πρόθεση της παιδείας στα μέσα και τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες και μπορούμε να επανέλθουμε στη συνέχεια όταν έρθει και η στιγμή για ερωτήσεις. Και τώρα... Μπορούμε να ακούσουμε κάποιες ε, ερωτήσεις ε, και απαντήσεις και μετά να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Έχουμε 20 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στον τρίτο μιλητή και στον εισηγητή μας. Λοιπόν, ο κύριος Στρασνογεύσκη, Στρογεύσκη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω κάποιες επικριτικές παρατηρήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η σημερινή συζήτηση για τις βιβλιοθήκες διεξάγεται με βάση τα όσα προβλέπουν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις ε, και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στις συγκεκριμένες πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης νέων μεγάλων βιβλιοθηκών. Ε, στα προηγούμενα πολιτικά σχέδια υπήρχε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τώρα, βάσει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μεγάλε βιβλιοθήκε ή κρατικά αρχεία. Δεύτερον, η συζήτηση αυτή γίνεται σε μια πολύ σημαντική ε, χρονική συγκυρία για την φορολόγηση των βιβλίων, των ηλεκτρονικών βιβλίων και των οπτικοακουστικών βιβλίων. Υπάρχουν ε, πολύ χαμηλοί φόροι στα βιβλία, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος για τη φορολόγηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Ε, τα νέα αυτά βιβλία, τα οποία βελτιώνουν τις δεξιότητες των πολιτών με χαμηλό κόστος. Αυτά τα δύο στοιχεία τα αναφέρω, διότι εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού μπορούμε να κάνουμε υποδείξεις και να ε, εκφράζουμε και τις επιθυμίες μας. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια εξαίρεση για τις βιβλιοθήκες και να ε, υποδείξουμε ποια είναι ε, τα ευρωπαϊκά μέσα τα οποία ναι μεν είναι βοηθητικά, δεν είναι κύρια, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν για τη χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών. Διότι αν αυτές οι μεγάλες βιβλιοθήκες που μας δείξατε εσείς στις διαφάνειές σας έχουν προκύψει από πολύ σημαντική χρηματοδότηση και αποτελούν πρέσβεις της ανάγνωσης. Στα ηλεκτρονικά βιβλία η υψηλή φορολόγηση θα δυσκολεύει την πρόσβαση τρίτη πρόταση και από εκεί και πέρα θα μπορούσα ίσως να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε, ε, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ποικίλα στατιστικά στοιχεία για την ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες και δεν είναι πάντα συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία. Σε πολλές ε, χώρες υπάρχουν στρατηγικά προγράμματα για την ανάγνωση, για την συμμετοχή σε προγράμματα τα οποία πολύ συχνά σχετίζονται και με εθνικά προγράμματα χρησιμοποιούμε μία ε, μέθοδο τελείως διαφοροποιημένη. Επομένως, το να λέμε τι γίνεται στη Σουηδία ή στη Δανία ή τι συμβαίνει στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία οδηγεί σε κάποιε αντιφάσει, γιατί ξεκινούμε από τελείω διαφορετική βάση αναφορά. Η προσωπική μου εμπειρία ως Υπουργό Πολιτισμού ε, με οδηγεί ε, στο εξή συμπέρασμα για την οργάνωση μιας βιβλιοθήκης, ο βασικός εταίρος για διάλογο δεν είναι ο Υπουργό Πολιτισμού, πολύ συχνά είναι ο Υπουργό Οικονομικών. Και εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, ιδίως ε, όσον αφορά αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε σήμερα. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά τα στοιχεία που μας δώσετε για τον Καναδά, ότι ένα δολάριο Καναδά ε, πολλαπλασιάζεται στην πραγματικότητα. Το ξέρει κάθε Υπουργό Πολιτισμού, αλλά κανένα Υπουργό Οικονομικών. Επομένω, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, παρουσιάσουμε. Πρέπει να δώσουμε κάποια παραδείγματα, να εξηγήσουμε πώ έχουν τα πράγματα στην αρχή. Οι ερωτήσει μου λοιπόν αφορούν σε αυτέ τι δύο παρατηρήσει που έκανα. Πώ έχουν τα στατιστικά στοιχεία για τι χώρε μέλη σε δυναμικό επίπεδο και πώ μπορούμε να αιτιολογήσουμε λίγο καλύτερα την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που δαπανούν για τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο στον πρώην Υπουργό Πολιτισμού της Πολωνίας, αλλά θα ήθελα να ζητήσω στους συναδέλφους να τηρήσουν ε, το χρονικό περιθώριο, 1,5 λεπτό το πολύ, 2. Η κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι για άλλη μια φορά οι δημόσιες βιβλιοθήκες διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο και βοηθούν και τις κοινότητες, βοηθούν την εκμάθηση της ανάγνωσης ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικές διότι προσφέρουν πρόσβαση σε πολλούς ανθρώπους και χρειάζεται κατεπηγόντω η βοήθειά του. Αναφερθήκατε στη συνέχεια στον εξυγχρονισμό των βιβλιοθηκών και θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Εσεί στο Διεθνή Οργανισμό σα συζητάτε το ερώτημα πού θα πρέπει να βρίσκεται αυτό το ταμείο και εάν υπάρχει καμία δυνατότητα από τι οργανώσει των Ευρωπαϊκών Βιβλιοθηκών να κάνουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το περιβόητο σχέδιο Juncker. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Γραμματικάκη είναι πολύ ωραία η σημερινή συνάντηση κυρία Πρόεδρε και τονίζει το ρόλο των βιβλιοθηκών. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ένας φανατικός φίλος, σχεδόν μανιακός, των βιβλιοθηκών και ένας με μεγάλες επιφυλάξεις φίλος ε, του διαδικτύου. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Αν κοιτάξετε την ανθρώπινη ιστορία, οι βιβλιοθήκες έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Αφιβάλλω πάρα πολύ για τα υπόλοιπα σύγχρονα μέσα τι ρόλο θα παίξουν. Και θα σας πω ένα καλό νέο. Από χορηγία ενός διάσημου αφοπλιστού σε έξι μήνες περίπου μια από τις καλύτερες βιβλιοθήκες της Ευρώπης θα είναι σε ένα ιστορικό μέρος στην Αθήνα. Οπότε θα περιλάβετε στις φωτογραφίες σας, σας παρακαλώ, και αυτή την καινούργια βιβλιοθήκη. Εθνική βιβλιοθήκη που δείχνει ότι ευτυχώς ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Και μια ερώτηση. Θα σας φανεί αφελής η ερώτηση. Αλλά δεν είναι. Και μάλιστα την υπέβαλα και στο διευθυντή της δικής μας βιβλιοθήκης, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και αυτός δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Ενώ τις πραγματικές βιβλιοθήκες και όχι τις ιντερνετικές βιβλιοθήκες. Ποιος, πώς και με ποια κριτήρια επιλέγει ποια βιβλία θα τοποθετηθούν στις βιβλιοθήκες φαντάζομαι όχι το καθένα που εκδίδεται, κάποιος τρόπος θα υπάρξει και προσέξτε την απάντησή σας γιατί είναι και λίγο παγίδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου τον Είστε πολύ ειλικρινείς. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Α, παρακαλώ. Ο κύριος Μαρακάλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα Ισπανικά αν επιτρέπετε. Εγώ ε, είμαι απόλυτα πεπισμένο για αυτά που μόλις εξηγήσατε, συμφωνώ απολύτως, επομένω η ερώτησή μου και αυτά που ζητάτε εσείς όσον αφορά τα κίνητρα είναι σχεδόν ε, ρητορικά. Γιατί να μην πάμε παραπέρα. Αυτά τα οποία εξηγήσετε και αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, που κάτι είναι και αυτό, είναι ότι το ζεύγος δημόσια βιβλιοθήκη σχολείο είναι μια βασική έννοια και είναι πρωτίστως σε μεγά... μικρότερες πόλεις ή σε χωριά και θα ήταν ακόμα καλύτερο εάν καταφέρναμε να ε, εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της ε, τεχνολογίας της πληροφορίας, όπως πολύ συχνά ακούσαμε σήμερα. Όμως, το πρόβλημά μας δεν είναι η ενημέρωση και η πληροφορία αυτή τη στιγμή, αλλά η κατανόηση. Το πρόβλημά μας είναι η ικανότητα να ερμηνεύουμε και να μην χαθούμε στον κικαιώνα των πληροφοριών που έχουμε από τις κοινωνίες μας και των προβλημάτων μας. Εγώ νομίζω ότι οι βιβλιοθήκες λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να αναλαμβάνουν την ευθύνη όχι μόνο να υποδέχονται ή να παρέχουν πρόσβαση ή να έχουν σύνδεση με σχολεία ή άλλα ιδρύματα, και όχι αυτή την ε, καταπληκτική αναφορά στην ε, αστική αξία της ε, βιβλιοθήκης, στην οποία και εγώ συμμετέχω και υποστηρίζω ακράδαντα. Πρέπει να αναφερόμαστε σε ανοιχτές πόρτες, αλλά να κάνουμε και κάτι πιο δραστήριο, πιο ενεργό. Να περάσουμε από την, το έργο της υποδοχής στο έργο της καθοδήγησης. Πιστεύω ότι η δημόσια βιβλιοθήκη θα πρέπει ε, να ε, ανταγωνίζεται ε, στα πλαίσια του εξαγωνίζεστε με τα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες που πραγματικά χρειάζονται αυτή την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προέλθει από τις βιβλιοθήκες. Από πληροφορίες ε, έχουμε. Να φάνε και κότες. Αλλά υπάρχουν και όλα αυτά τα περίπλογα στοιχεία και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε καταλήλως. Αυτό λοιπόν το οποίο σας ζητώ είναι εάν απέχουμε ή αν πλησιάζουμε να δώσουμε αυτό το επιπλέον βήμα για έναν ακόμα ρόλο για τις βιβλιοθήκες ε, και τη σχέση τους με τα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. E altri? No. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις, αν με επιτρέπετε. Η πρώτη είναι εξή. Όσον αφορά τους σπόρους που ανέφερε και ο συνάδελφος Δρογέσκη. Νομίζω ότι και από αυτό το ενδιαφέρον έγγραφο που έχουμε ζητάτε πρόσβαση σε πόρους και ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα ήθελα να ξέρω σε ποια προγράμματα συμμετέχετε ήδη, μπορείτε να συμμετέχετε, διότι και ως ε, Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία νομίζω ότι έχετε πρόσβαση σε κάποια προγράμματα, στο Erasmus Plus για παράδειγμα. Ε, δεν ξέρω όμως αν συμμετέχετε για παράδειγμα σε όλα αυτά τα προγράμματα, γιατί εμείς δώσαμε μεγάλη μάχη για να περιλαμβάνεται ο πολιτισμός ε, και ε, η ψηφιακή ε, τεχνολογία και να συμμετέχετε και σε αυτά τα προγράμματα τα οποία δεν δίνουν χρηματοδότηση για τις δομές αλλά δίνουν για παράδειγμα για την κατασκευή πλατφόρμας. Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά, εάν δεν θυμάμαι λάθος, υπάρχει ένα ανώτατο όριο 5 ε, εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν υπήρχε. Αυτό αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία. Βέβαια θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στο σημείο αυτό. Και βεβαίως για τα διαρθρωτικά ταμεία ε, υπάρχει χρηματοδότηση μόνο εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να καταλάβω λίγο καλύτερα. Όταν λέτε χρειαζόμαστε πόρους για την καινοτομία, δεν αφορά μόνο την ψηφιακή καινοτομία, αλλά φαντάζομαι ότι αφορά και άλλη μορφή καινοτομία. Δεύτερον, στι προτάσει σα, ε, τι οποίε ε, είδα στο έγγραφό σα, μία από τι ενδιαφέρουσε προτάσει είναι να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σήμα. Ένα ευρωπαϊκό σήμα βιβλιοθηκών. Θα αναφερθούμε φυσικά σε πρότυπα, σε αναγνώριση του ρόλου των βιβλιοθηκών. Αυτά θα ήθελα να τα καταλάβω λίγο καλύτερα για τις ε, ψηφιακές γνώσεις και τις ψηφιακές δεξιότητες Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέσεις ε, με τα δίκτυα των σχολικών βιβλιοθηκών. Είναι εθνικά αμυγός ή υπάρχουν κάποιες συστάσεις άλλες. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτή η πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνετε, με την οποία συμφωνώ, είναι ότι η προσέγγιση της UNESCO προβάλλει περισσότερο τα πολιτιστικά στοιχεία. Μήπως υπερβάλλουμε λοιπόν ε, στην ε, ψηφιακή και τεχνολογική προσέγγιση και όσον αφορά τις διαξιότητες αλλά και όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των βιβλιοθηκών. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε εσείς κάποιες ιδέες από αυτό γιατί εμείς πολύ θα θέλαμε να συμμετέχουμε, να βοηθήσουμε και να διορθώσουμε αν χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσετε τώρα και στη συνέχεια θα περάσουμε... Α, θέλετε να δώσετε το λόγο προς τους ε, αυτούς... Ο κύριος Βέντα και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μία απλή ερώτηση έχω. Μετά από αυτές τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις και τα λέγες απόψεως πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα πολύ καλό μήνυμα. Έχουμε 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Δεν το ήξερα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ποιες είναι οι τάσεις όμως, είναι αυξητικές οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε ορισμένες περιφέρειες. Ποιες λοιπόν είναι οι τάσεις, εκεί υπάρχουν αυξητικές τάσεις ή οι δημόσιες βιβλιοθήκες ψάχνουν νέους τρόπους συνεργασίας. Ε, ποια είναι τα δεδομένα που έχουν ενδεχομένως αλλάξει σχέση με 10 χρόνια πριν. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλετε να απαντήσετε. Well, Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε με το χρήμα πρώτα. Ερωτήσατε κάποιοι για το αν οι δημόσιες βιβλιοθήκες συμμετέχουν σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει γίνει ήδη αυτό στη δεκαετία του 90. Υπήρχε το πρόγραμμα «Publica» τότε, το οποίο βασιζόταν στην καινοτομία ε, στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Αυτό ήταν κάτι καινούργιο και ε, πολλές βιβλιοθήκες επωφελήθηκαν και προχώρησαν, εξελίχθηκαν. Εξελίχθηκαν και οι ιδέες ε, για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια βιβλιοθήκη. Κάποιες μεμονωμένες βιβλιοθήκες έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω των τοπικών τους κυβερνήσεων. Αγοράστηκαν, για παράδειγμα, λεωφορεία που μετατράπηκαν σε κινητές βιβλιοθήκες έγιναν ανακαινήσει, όμως αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά για ε, μεμονωμένε βιβλιοθήκες. Δεν υπάρχει δηλαδή μια γενικευμένη κατάσταση. Εξαρτάται από τις τοπικές αρχές και πολλές φορές οι τοπικές αρχές έχουν άλλες προτεραιότητες και δεν φτάνουν τα χρήματα λοιπόν σε μια βιβλιοθήκη. Τώρα, νομίζω ότι Ούτε στη Γερμανία, σίγουρα όχι στη Γερμανία, ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Εμείς αυτό που προσπαθούμε μέσω των ε, διαφόρων ευρωπαϊκών ε, οργανισμών να βρούμε χρηματοδότηση για να στηρίξουμε αυτές τις στατιστικές. Όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικά τα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα κυρίως που ε, μαθαίνουμε για το τι συμβαίνει στις βιβλιοθήκες. Είναι λοιπόν σίγουρα κάτι σημαντικό και αυτό έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 90, όμως τότε χρησιμοποίησαμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν ε, μας έδωσαν άλλη χρηματοδότηση. Ε, τώρα, θετικές τάσεις. Παιδιά σίγουρα υπάρχουν παντού. Παιδιά που έρχονται με τους πρόσφυγες, τα οποία αυξάνονται οι δημόσιες βιβλιοθήκες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να μάθουν σε ένα χώρο διαφορετικό από ό,τι στο σχολείο. Ε, και ο κύριος Γραμματικάκης ε, μας ρώτησε γιατί να υπάρχει κτίριο όταν υπάρχει το διαδίκτυο. Να σας απαντήσω. Υπάρχει το κτίριο φυσική βιβλιοθήκη διότι εκεί βρίσκεται ένα σύνολο πολιτισμού πληροφοριών. Υπάρχει μια ωραία μίξη και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που δεν έχει αμυγός εκπαιδευτικό χαρακτήρα διότι η βιβλιοθήκη δεν είναι εκπαιδευτικό ε, οργανισμός όμως είναι ένας χώρος μάθησης και πιστεύω πως αυτοί οι χώροι μάθησης θα γίνουν ε, πιο σημαντικοί. Ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνει το παιδί και συνειδητοποιεί ότι αφού τελειώσει το σχολείο υπάρχει ένα μέρος που μπορεί να πάει σε αυτό και να συνεχίσει να μαθαίνει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, αυτό που μας είπατε με την Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Νιάκου στην Αθήνα και με χαρά μου να έρθω και να την επισκεφτώ. Ε, να συνεχίσω τις απαντήσεις μου. Όχι, εσύ συνάδελφα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις ερωτήσεις. Ε, κύριε Γραμματικάκη, η ερώτησή σας για το αν χρειάζεται μια βιβλιοθήκη, το κτίριο μιας βιβλιοθήκης πλέον. Να σας αναφέρω δύο πράγματα. Καταρχάς, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε έχει σταθεροποιηθεί. Βλέπουμε ότι ε, σταθερά μειώνεται. Είναι ε, το 30% της αγοράς βιβλίου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, το 70% όλων των βιβλίων που ε, πολλούνται είναι ε, βιβλία όχι ηλεκτρονικά, είναι έντυπα. και ένα αντίστοιχο ε, ποσοστό ανθρώπων όταν ερωτήθηκαν αν προτιμούν να διαβάζουν από ένα έντυπο βιβλίο ή από την οθόνη ε, μας απάντησαν ότι προτιμούν να διαβάζουν το χάρτινο βιβλίο, την έντυπη έκδοση. Αυτό ισχύει και για τα παιδικά βιβλία. Ρωτήσαμε παιδιά, νέους αναγνώστες και μας είπαν ότι προτιμούν να διαβάζουν από χαρτί τώρα πολλοί φοιτητέ, ε, σπουδαστές, οι οποίοι έχουν ψηφιακή διδακτέα ύλη, πολλές φορές προτιμούν να εκτυπώνουν αυτήν την ύλη και να τη διαβάζουν από χαρτί. Είναι λοιπόν εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αφού ε, έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλά πράγματα αυτό θα ισχύσει και για τα βιβλία. Όμως στην περίπτωση αυτή νομίζω πως ε, δεν ισχύει αυτό. Επίσης, είναι προτιμότερο φυσικά να ε, παραμείνουμε στις έντυπες εκδόσεις, όχι μόνο στις δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά και γενικότερα. Επίσης, για να συνεχίσω την απάντησή μου ε, και στην ερώτηση του κυρίου Μαραγκάλ. Θα μπορούσαν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, οι βιβλιοθήκες να είναι πιο ενεργές και να προσπαθήσουν να συμμετέχουν περισσότερο στις ε, τοπικές κοινωνίες. Να σας πω πώς εξαρτάται από το που βρίσκεται κανείς. Για τη δική μου χώρα, για τις κάτω χώρες, μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Βιβλιοθήκη στα σχολεία. Είναι ένα πρόγραμμα που έχουν διοργανώσει δημόσιες βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν κάποιες ε, δυνατότητες δανεισμού στα σχολεία. Υπάρχει δηλαδή μία βιβλιοθήκη, σχολική βιβλιοθήκη, την οποία διαχειρίζεται η δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα σχολείο ή μπορεί κάποιος ε, να ψάξει στους υπολογιστέ να ζητήσει κάποια βιβλία, να τα δανειστεί από τη βιβλιοθήκη η οποία με τη σειρά τη θα τα φέρει στα σχολεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Διαχειρίζεται δηλαδή η εκάστοτε τοπική δημοτική αρχή το πρόγραμμα αυτό. Και αυτό γίνεται συνήθως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν στο σχολείο δεν υπάρχει κάποια δανειστική βιβλιοθήκη, οργανωμένη από τις ε, δημόσιες βιβλιοθήκες, τότε η βιβλιοθήκη που έχει το ίδιο το σχολείο είναι κατώτερης ποιότητας. Και σίγουρα λοιπόν οι δημόσιες βιβλιοθήκες προσπαθούν να συνεργαστούν με τα σχολεία, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα και σε άλλους τομείς. Σίγουρα όμως ε, πρέπει να προσέξουμε να μην επιδεινωθεί και το επίπεδο των ε, δανειστικών βιβλιοθηκών στα σχολεία, όπως έχει συμβεί στις κατοχώρες. Τώρα, στατιστικά στοιχεία. Ναι, εγώ προσωπικά προσπαθώ εδώ και 10 χρόνια να συγκεντρώσω στατιστικά στοιχεία τα οποία θα είναι αξιόπιστα, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να τα αξιολογήσουμε. Και μιλώντας για κίνητρα, σίγουρα χρειάζεται να δοθούν κίνητρα από κάποια υπερεθνική οντότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορούν να συλλέγονται αυτά τα στατιστικά στοιχεία με καλύτερο τρόπο στο μέλλον για ε, να δούμε κι εμείς πώς θα κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Ή μπορεί οι στατιστικές υπηρεσίες να μας βοηθήσουν για αυτό το σκοπό. Και θα ήταν καλό. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και δεν έχουμε ε, όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μας. Τώρα, για να ολοκληρώσω αυτός ο γραμματισμός που αναφέρατε στα ψηφιακά μέσα. Αν κατάλαβα καλά αυτό που με ρωτήσατε, ε, σχετίζεται περισσότερο με το πρόγραμμα της UNESCO. Και δεν είναι τόσο τεχνικό το ζήτημα, σωστά. Όχι, σύμφωνο και εγώ μαζί σας. χρειάζεται να προσανατολιστούμε περισσότερο στην πολιτισμική πτυχή και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό είπα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να έχουμε επίγνωση όλων των πτυχών του ψηφιακού γραμματισμού και των πιο ήπιων Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να ερμηνεύουμε ε, όλες ε, τις ε, πληροφορίες και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτές. Να δούμε γιατί ας πούμε έχουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία, ποιος την έχει στείλει, για ποιο λόγο. Σας ευχαριστώ. Sorry, we have another Υπάρχει και άλλος ομιλητής. Δεν μπορείτε να ρωτήσετε μετά. Δεν είναι ερώτηση. Δεν είπα ποτέ ότι εγώ είμαι εχθρός της δημόσιας βιβλιοθήκης. Είπα το αντίθετο ακριβώς. Ναι, είπατε προηγουμένως ότι αγαπάτε πολύ τις βιβλιοθήκες. Παρακαλώ. Να δώσω το λόγο στον τρίτο και τελευταίο ομιλητή για ειδικό για την ε, ψηφιακή και διαδικτυακή πολιτική, τον κύριο Νταν Μούντ. Για τον ηλεκτρονικό δανεισμό. Θα μπορούσατε να απαντήσετε και για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Okay. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να ακολουθήσω ε, την Μπάρμπαρα και τον Φράνξε. Έκαναν εξαιρετικές παρουσιάσεις ε, για τα δικά τους θέματα. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με, την, ε, τον ηλεκτρονικό δανεισμό. Ε, υπάρχει δομή μέσα στο έγγραφό μου, βάζω και τη σωστή διαφάνεια. Θα ήθελα να πω στην αρχή της παρουσίασής μου πως ε, καλό είναι να δούμε ιστορικά την πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες. Όσο επιτοπλίστων στην ιστορία η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα πολιτιστικά προϊόντα και στις γνώσεις ε, ήταν πραγματικά πλεονέκτημα μόνο για τους λίγους και εκλεκτούς. Τα τελευταία 200 ε, χρόνια μπορούμε να πούμε μετά την βιομηχανική επανάσταση και την εξάπλωση των προγραμμάτων αλφαβητισμού και γραμματισμού κυρίως στις είπα είδαμε μια ε, διαφορετική πορεία και υπάρχουν πλέον φορεί ε, που προωθούν την πρόσβαση στην ε, εκμάθηση, στις γνώσεις, στα πολιτιστικά προϊόντα και δημιουργούνται και φυσικά και κίνητρα για τους πνευματικούς δημιουργούς. Ε, μιλώντας για τον δανεισμό των βιβλίων, πολλά καθεστώτα υπάρχουν σε χώρες ε, για να μπορέσουν ε, να ε, προβούν σε δανεισμό με την κατάλληλη αποζημίωση φορείς. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια επανάσταση με αυτήν την εξέλιξη και αυτό οδήγησε σε αλλαγές ως προς τους εκδοτικούς οίκους και τις δημοτικές βιβλιοθήκες και βλέπουμε ότι σταδιακά η άδεια για πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο περιεχόμενο αντικαθιστά την κατοχή του βιβλίου. Όταν κατεβάζετε ένα βιβλίο ή ένα τραγούδι ή οτιδήποτε στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σα. δεν το κατέχετε, έχετε απλώ την άδεια για πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και έχετε ε, ε, συμφωνήσει με του όρου χρήση. προτού σα χορηγηθεί η άδεια χρήσης. Μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι είστε κάτοχος, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικέ ε, διαφορέ και κυρίω για τι δημόσιε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι μεγάλη μεγάλη πρόκληση, διότι δεν υπάρχει η ίδια νομική βάση για τον δανεισμό που σας έλεγα προηγουμένως, οπότε πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους εκδοτικούς οίκους αμέσα για να έχουν την άδεια πρόσβασης και να μπορέσουν δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να δανείζουν ψηφιακά τα βιβλία. Ως αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες ανέπτυξαν διάφορα είδη αδειών. Ναι, θα ε, ανατρέξω σε πέντε βασικές κατηγορίες. Πρώτον, ε, το μοντέλο του ε, νέου χρήση, δηλαδή μία άδεια ανά χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουν εξαντληθεί οι άδειες, τότε θα πρέπει να περιμένετε για να... μια ηλεκτρονική λίστα αναμονής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδοσιακές τριβές, όπως και για το δανεισμό των βιβλίων όμως ε, για τις βιβλιοθήκες ε, βλέπουμε ότι είναι τεχνητά περιοριστική αυτή η όρη διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα καταναλωτικά μας πρότυπα στη ψηφιακή κοινωνία. Το υβριδικό μοντέλο δανεισμού είναι ένας συνδυασμός διαφόρων προτύπων αδειών, ε, άδεια αναχρήστη, άδεια ταυτόχρονης χρήσης ε, και άδεια συγκεκριμένης διάρκεια, εξάμηνη παραδείγματο χάρη και πρέπει να ανανεωθεί όταν εκπνεύσει και είναι συνδυασμός αυτών των ε, τριών διαφορετικών αδειών με διαφορετική τιμολόγηση. Ποιο είναι το πλεονέκτημα. Υπάρχει η μεγαλύτερη επιλογή, μεγαλύτερη ευελιξία για τις βιβλιοθήκε, αλλά ε, αυτό επισύρει και μεγαλύτερο κόστο και περιπλοκότητα ε, για αυτέ και για του χρήστες. Για την άδεια των βιβλιοθηκών που ε, καταβάλλεται αποζημίωση στον εκδοτικό οίκο από την βιβλιοθήκη. Αυτή είναι, αυτό είναι το πιο σύνθεσμο μοντέλο, αλλά δεν περιορίζεται ο ρυθμός των ταυτόχρονων χρηστών. Όμως, ε, αν ε, εκατοντάδες χιλιάδες θέλουν να δανειστούν αυτό το βιβλίο, τότε θα υπάρχει ένα πρόβλημα με τις πληρωμές προς τον εκδοτικό οίκο. Δεν θα το σηκώσει το σύστημα, αν θέλετε, και όταν υπάρχουν σημεία εχμής ως προς τη ζήτηση, τότε ε, δημιουργείται ε, πρόβλημα και δεν μπορεί κάποιος να δανειστεί τη βάση αυτού του μοντέλου το, το βιβλίο που επιθυμεί. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας για τα καταναλωτικά πρότυπα μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ναι. Το δεύτερο μοντέλο, η διτή άδεια, ε, στη Δανία και στη Σουηδία χρησιμοποιείται από τα 18 μοντέλα δηλαδή που εξέτασα εγώ ε, αυτό προέκυψε και οι δημόσιες βιβλιοθήκες συνδέονται με τους εκδοτικούς οίκους και υπάρχει η ψηφιοποίηση από πλευράς των εκδοτικών οίκων ε, και παρέχεται και εκδοτικό δικαίωμα προς τις βιβλιοθήκες δηλαδή είναι win-win situation ε, βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε περιορισμένες αγορές για μικρές γλώσσες, ε, ενώ για τα αγγλικά παραδείγματο χάρη ε, οι οικονομίες ε, κλίμακας επιτρέπουν την ψηφιοποίηση για τους ίδιους εκδοτικούς οίκους χωρίς να χρειάζεται να παρεμβαίνουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες για τέτοια πράγματα. Ε, τέλος, το μοντέλο των δημοσίων βιβλιοθηκών που συνεπάγεται κατοχή ψηφιακής υποδομής, ε, δηλαδή λειτουργεί ως σερβερ, ως σημείο αποθήκευσης η βιβλιοθήκη για όλο το ψηφιακό περιεχόμενο. Ε, σε κατά αντιδιαστολή με τα προηγούμενα μοντέλα που βασιζόμαστε σε εξωτερικούς διαμεσολαβητές για τον ψηφιακό δανεισμό ε, και επιπροσθέτως συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και η δημόσια βιβλιοθήκη, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν τρίτη φορείς που είναι απαραίτητοι και πλατφόρμες τους να για τον δανεισμό. Λοιπόν, σε αυτό το μοντέλο η δημόσια βιβλιοθήκη αποθηκεύει το περιεχόμενο και σε ε, ε, ψηφιακούς όρους δεν υπάρχει μεγαλύτερο δικαίωμα κατοχής, ε, ιδιοκτησίας αν θέλετε και η διαδικασία δανεισμού ελέγχεται από την ίδια τη δημόσια βιβλιοθήκη. Ποιο είναι το μειονέκτημα, χρειάζονται υψηλότατες επενδύσεις και για την δημιουργία αυτού του συστήματος αλλά και για την εξάπλωσή του όσο προστίθενται νέοι τίτλοι. Οι δημόσιε βιβλιοθήκες δεν έχουν στόχο να προσφέρουν φυσικά του πλέον δημοφιλεί τίτλου, για προφανεί ε, λόγου, οπότε μπορούμε να δούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πέρα από αυτό τη σύγκριση των διαφόρων μοντέλων ε, μπορώ να σας πω ότι από Κατέληξα ε, στο εξή ε, συμπέρασμα ότι το, ο ψηφιακός δανεισμός αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό δανεισμού, δηλαδή από 1 έως 10% ανάλογα με τη χώρα. Πάντως μειώνεται το ποσοστό ε, του δανεισμού βιβλίων και αυξάνεται ραγδαία το ποσοστό του ψηφιακού δανεισμού. Για το 2005 παραδείγματος χάρη είχαμε 100 20 εκατομμύρια σε σχέση, δηλαδή αύξηση από τα 75 εκατομμύρια το 2014 ε, και αντίστοιχα ε, μειώθηκε δηλαδή ο δανεισμός των βιβλιοσικών βιβλίων και τα, αυξήθηκε αντίστοιχα από τα 2,9 στα 3,8 εκατομμύρια ο ψηφιακός δανεισμός ε, για την ίδια περίοδο. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα σημεία σύγκρισης. Ε, ε, θέλω βεβαίως να συνειδητοποιήσετε ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες πίσω από κάθε ρυθμό και ποσοστό που βλέπετε. Παραδείγματο χάρη για το υβριδικό μοντέλο Σλοβενία βλέπουμε πως μπόρεσαν το 8% των διαθέσιμων ηλεκτρονικών βιβλίων να καταστούν διαθέσιμα στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Είναι σημαντικό αυτό το επίτευγμα. Αλλά αυτό αντιστοιχεί σε 800 τίτλους από τους χίλιους που υπήρχαν το 2014. Ε, αντίθετα, όταν βλέπουμε για την Ουαλία τι συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά βιβλία, ε, έχουν το 0,7% απογοητευτικό ποσοστό για, τις, ε, για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Όμως, αυτό έχει σε 12.000 τίτλους, πολύ περισσότερους επειδή είναι τόσο μεγάλη αγορά των ε, αγγλόφωνων βιβλίων. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να αξιολογήσετε αυτά τα, αυτά τα ποσοστά λαμβάνοντας υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες. Ε, επίσης, για τα μοντέλα του ηλεκτρονικού ψηφιακού δανεισμού, ε, κυρίως στην Αμερική, αυτά που εξέδεσα, βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, ως προς τις πολιτικές που ακολουθούνται για την πρόθεσή τους μέσα από τοπικά πιλωτικά προγράμματα ή αντίθετα ε, μέσα από εθνικές πολιτικές για την αδειοδότηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι τα ο πολιτιστικός παράγοντας. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, ε, το μοντέλο ηλεκτρονικού δανεισμού ε, ε, εποφελείται από το EKZ τι είναι αυτό, είναι η Κεντρική Ένωση για τα, την αγορά βιβλίων ε, δημόσιας χρήσης. Αν θέλετε, η αποθήκη των ε, δημοσίων βιβλιοθηκών ε, προσφέρουν υπηρεσίες, έπιπλα και ούτω καθεξής. Έχουν πάγια σχέση λοιπόν με τις δημόσιες βιβλιοθήκες και γενικά είναι αποδεκτό ότι η απογείωση του μοντέλου του ηλεκτρονικού δανεισμού στην Γερμανία τα τελευταία χρόνια μπορεί να αποδοθεί και στην ύπαρξη αυτής της ε, υποδομής. Ε, επίσης, ε, εκπρόσωποι φορέων ηλεκτρονικού δανεισμού στο Κεμπέκ μου είπαν ότι έχουν πολύ ψηλά ποσοστά διότι ιστορικά υπήρχε πολύ σημαντική συνεργασία με τις βιβλιοθήκες. Δηλαδή ε, αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι οι, δημοσια... οι δημόσιες βιβλιοθήκες ε, δεν ακολουθούν την εμπορική αξία του βιβλίου για να παραγγείλουν ε, τα βιβλία τους και νομίζω ότι αυτός ο ρόλος των δημοσίων βιβλιοθηκών μπορεί να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό δανεισμό σε πολλές χώρες. Τρέχω λίγο γιατί δεν έχω χρόνο. Ε, νομίζω ότι για την παροχή της υπηρεσίας, τη διατήρηση και της εξάπλωσης είναι σημαντικό να δώσουμε και την δόση σημασία στις διαπραγματεύσεις. Ε, μπορεί να υπάρχουν πολλά προβλήματα με την συμπεριφορά των εκδοτικών οίκων, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η διαθεσιμότητα των τίτλων σε ε, μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Θα επανέλθω σε αυτό σε γιατί δεν έχω χρόνο τώρα. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο στα συμπεράσματά μου. Υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα, διάφορες συστάσεις. Ε, ε, δεν μπορούμε να επιδιώξουμε ένα ενιαίο μοντέλο, κατά τη γνώμη μου. Αυτή την ε, συγκριτική μελέτη που έκανα για όλες αυτές τις χώρες, για τα 18 διαφορετικά μοντέλα, βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση, οι πολιτιστικές προσδοκίες και τα ιστορικά πρότυπα οδηγούν σε διαφορετική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού δανεισμού. Δηλαδή, υπάρχουν, μπορούμε να αντλήσουμε δάγματα από κάθε διαφορετικό μοντέλο, ας τα ε, ε, προσεγγίσουμε ως ε, μικρά εργαστήρια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πάρω ένα από αυτά τα 18 μοντέλα και να το προτείνω ως ιδανικό για όλους. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό αυτό. Τι πρέπει να γίνει τώρα για τις δημόσιες βιβλιοθήκες και για τους εκδοτικούς οίκους, επειδή όλοι έχουν ιδεατούς στόχους οποίους επιδιώκουν, θα πρέπει να τονίσω ότι μετά την συγκριτική μελέτη που έκανα, καταλήγω στο ότι χρειάζονται συγκεκριμένα μικρά βηματάκια κάθε φορά για να μπορέσουμε τελικά να υλοποιήσουμε τους μεγαλεπίβολους στόχους μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βασιζόμαστε σε αμοιβαία κατανόηση ανταλλαγή πληροφοριών και νομίζω ότι αυτό τονίστηκε. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα για δημόσιες βιβλιοθήκες. Ε, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε σημεία σύγκριση ε, σε συγκριτικό επίπεδο για το δανεισμό. Δηλαδή χρειάζεται μια χαρτογράφηση τη της πραγματικότητας ως προς τη συμπεριφορά των χρηστών αλλά και των δημόσιων βιβλιοθήκων βιβλιοθηκών σε σχέση με την εμπορική αξία των βιβλίων για να βελτιώσουμε τις σχέσεις και τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι δημόσιες βιβλιοθήκες και οι εκδοτικοί. Δηλαδή όταν δεν έχουμε τις γνώσεις ε, κυρίως αποφεύγουμε τον κίνδυνο. Ε, αυτή είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά και το ίδιο κάνουν και οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Αν υπάρχουν λοιπόν ε, περισσότερες γνώσεις θα επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία, ώστε με ευελιξία να σχεδιαστεί η πολιτική δανεισμού και να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα περιορισμένα ομολογουμένω κονδύλια που υπάρχουν. Μπορούμε να, διερευνήσουμε και άλλου τρόπους για εξάπλωση, διεύρυνση του μοντέλου δανεισμού σε σχέση με τα εφιστάμενα εμπορικά μοντέλα. Ε, δεν έχω άλλο χρόνο όμω, θα σταματήσω εδώ και μετά τι ερωτήσει θα επανέλθω σε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που δεν έχει αμέσως σχέση με τον ηλεκτρονικό οργανισμό, αλλά με τρόμαξε μπορώ να πω. Αναφέρατε το παράδειγμα των κάτω χωρών, όπου ο οργανισμός βιβλίων έπεσε από 120 εκατομμύρια στα 75 εκατομμύρια. Αυτό δηλαδή Α, επίσης μας είπατε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία αυξήθηκαν από 2,9 στα 3,8. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο δανεισμός ε, έντυπων βιβλίων μειώθηκε και αυξήθηκε ο δανεισμός ηλεκτρονικών βιβλίων. Αυτό δηλαδή για μένα σημαίνει ότι ε, αυτή, αυτός ο ηλεκτρονικός δανεισμός δημιουργεί ανισορροπίες. Ε, υπάρχει κάποια στρατηγική, ή κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στη μείωση ε, που θεωρώ πως είναι δραματική του δανεισμού έντυπων βιβλίων. Θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις και μετά. Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο, πώς βλέπετε το δικό μας το ρόλο της ε, Επιτροπής μας ε, κατά την ανάπτυξη του ε, φαινομένου και της πρόσβασης των βιβλίων στο διαδίκτυο. Ο κύριος Μόργανο, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από την παρουσίαση είναι να δούμε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο τι λειτουργεί αμέσω. Το ερώτημα είναι μπορούμε να έχουμε μια υπόθεση μελέτης η οποία θα εξετάζει τις δυνατότητες της αγοράς με τον τομέα της παραγωγής ε, για να μπορέσουμε να έχουμε και κάτι το οποίο να είναι πιο στέρεο διότι θεωρώ ότι το όλο θέμα των βιβλιοθηκών ε, εκτός και αν υπάρχει μια εξαιρετική εξαίρεση όπου μπορεί να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση ε, υπάρχει θέμα οικονομικής βιωσιμότητας και από εκεί και πέρα εξυγχρονισμού και κατάλληλης πρικοδότησης. Εάν δεν υπάρχουν αυτά από κοινού και δεν μπορούμε να δούμε τι παραγωγή έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εντό αγωγικών και τη δυνατότητα πώληση όλων αυτών ε, τα οποία δεν είναι ε, το best seller για παράδειγμα, το πιο ευπόλυτο βιβλίο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τουλάχιστον όχι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Η κυρία Τρούπελ για την τελευταία ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του ηλεκτρονικού δανεισμού και τις διάφορες δυνατότητες που επισημάνετε για τα διάφορα μοντέλα διοδότησης και μας είπατε ότι ε, θέλουμε να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο θα διαπραγματευτούμε ώστε να βρούμε και τον καλύτερο τρόπο να το υλοποιήσουμε αυτό. Ξέρουμε όμως ότι κάποιοι εκδότες δεν είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν ακόμα. Θα ήθελα να θέσω και την εξή ερώτηση λοιπόν και προς εσάς αλλά και στους άλλους δύο μιλητές από τη Γερμανία και από την Ολλανδία. Εσείς πώς προσεγγίζετε το θέμα ε, ε νομοθετική λύση ή ε, μια διαπραγμάτευση και ένα διάλογος. Παρακαλώ. Νομίζω ότι θα απαντήσω τις ερωτήσεις ε, με αντίστροφη σειρά. Καταρχάς να απαντήσω στην ερώτηση της κυρία Στρούπελ για να εξοικονομήσουμε και χρόνο γιατί μακρηγόρησα λίγο παραπάνω από όσο περίμενα και δεν κατάφερα να αναφερθώ στη μεταρρύθμιση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως ε, με απόφασή του για την, ε, το νομικό καθεστώς της ηλεκτρονικού διανυσμού που αναμένεται βάση τη νομοδότησης που έχουμε είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια νομική βάση για τον ηλεκτρονικό δανεισμό βάσει συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει. Και αυτό ε, γίνεται και στα πλαίσια της αναθεώρησης των θεωμάτων ε, πνευματικών δικαιωμάτων και η Επιτροπή σας έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Τώρα, τα δικαιώματα δανεισμού, τα οποία αφορούν τον ηλεκτρονικό διανεισμό μπορεί να ισχύει και για τις βιβλιοθήκες, ώστε να νομιμοποιηθεί το ηλεκτρονικός διανεισμός και να υπάρχει και μια νομική βάση που να το καλύπτει αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν οι εκδότες εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο ηλεκτρονικός δανεισμός είναι απειλή για το επιχειρηματικό μοντέλο και πάλι θα χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα προκειμένου να αποθαρρύνουν ή να περιορίσουν τον ηλεκτρονικό δανεισμό και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε και τη γενικότερη εικόνα δέσμευσης και διαλόγου διότι αν αναζητούμε απλώς μια νομική λύση ε, δεν νομίζω ότι εν τέλει θα είναι ικανοποιητική. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και ε, να σχολιάσετε μάλλον εσείς πριν απαντήσω στις επόμενες ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη οι ε, συνεδρίες καθυστέρηση και πρέπει να φύγω πολύ σύντομα γιατί έχω ένα τρένο. Ε, η ερώτηση για τη Γερμανία και ε, τις λύσει τις οποίες ε, θα καταλήξουμε μετά από διαπραγμάτευση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι εκδότε δεν είναι πάντα διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν μαζί μα. Ορισμένε φορέ έχουν και νομικά προσκόμματα, όπω και εμεί. Υπάρχει όμως και το θέμα της δημιουργίας εμπιστοσύνης. Ο σύνδεσμος εκδοτών στη Γερμανία λέει ότι από νομική σκοπιά δεν μπορούν να διαπραγματευτούν με την Γερμανική Ένωση Βιβλιοθηκών γιατί αυτό είναι μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται ούτε βάσει εθνικού δικαίου ούτε βάσει κοινοτικού κεκτημένου που σημαίνει ότι όλες οι βιβλιοθήκες ε, ή οποιοδήποτε σύνδεσμος ή ένωση θα πρέπει να διαπραγματευτεί με κάθε εκδότη. Και είναι πάρα πολλοί εκδότες ακόμα στη Γερμανία, επομένως οι δημόσιες βιβλιοθήκες, έχουμε περίπου 2.000 δημόσιες βιβλιοθήκες στη Γερμανία, ε, πολύ κα άνετα θα μπορούσαν να δεχτούν να διαπραγματευτεί η Ένωση εκ μέρου όλων. Και αυτοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με του εκδότε, αν το επιθυμούν. Και υπάρχουν εκδότε οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται με το Σύλλογο, επομένω δεν έχουμε και τα προϊόντα των εκδόσεών του στι βιβλιοθήκε. Και νομίζω ότι ορισμένε φορέ είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα γιατί είναι αρκετά μεγάλοι εκδότε αυτοί είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το, πράγμα, ε, το πρόβλημα. Ε, η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι καλή. Εγώ είμαι υπέρ τη διαπραγμάτευση, αλλά ορισμένε φορέ δεν ε, λειτουργεί και δεν βοηθά το μέλλον. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για να προσθέσω κι εγώ κάτι. Νομίζω ότι η νομική λύση θα μπορούσε να βοηθήσει υπό την έννοια ότι η ισορροπία μεταξύ ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, η διαπραγμάτευση μεταξύ εκδοτών και βιβλιοθηκών μπορεί να είναι λίγο στρεβλή. Είναι τελείως διαφορετική η διαπραγμάτευση για τα ηλεκτρονικά βιβλία με τους εκδότες από ό,τι για τα έντυπα. Ε, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητά μια υπόθεση αυτή τη στιγμή ή μάλλον ζητήθηκε ε, γνωμοδότηση από Ολλανδό δικαστή για τα ε, δικαιώματα δημοσίου διαδανεισμού και κατά πόσο μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία σε αυτά τα δικαιώματα. Και προς έκπληξη αρκετών παρατηρητών και του υποφαινομένου, στην ε, προδικαστική απάντηση το δικαστήριο είπε ότι ε, ναι, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Εάν λοιπόν ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεκτεί τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα, μπορεί να επανέλθει η τάξη όπως ανέφερα προηγουμένως. Επομένως, τουλάχιστον οι δημόσιες βιβλιοθήκες θα έχουν το δικαίωμα να δανείσουν οποιοδήποτε βιβλίο, οποιοδήποτε τίτλο επιθυμούν. Ε, το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό λοιπόν είναι εν μέρη απάντηση στα όσα ρώτησε η κυρία Φερχάγεν. Εάν ε, τα συγκρίνετε αυτά όσον αφορά τα έντυπα βιβλία και τα ηλεκτρονικά βιβλία, δεν μπορείτε στην πραγματικότητα να κάνετε σύγκριση διότι πολλές από τις δικτυακές πύλες ηλεκτρονικού ε, δανεισμού έχουν περιορισμένο αριθμό τίτλων, επομένως δεν μπορεί να γίνουν πολύ δημοφιλείς όπως ε, ε, μια συλλογή μιας βιβλιοθήκης, όπου μπορούν να προσφέρουν οποιοδήποτε τίτλο να στην αγορά προς δανεισμό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Α, πρέπει να απαντήσετε και τις υπόλοιπες. Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε τελειώσει. Μάλιστα. Ε, αντίστροφη σειρά, όπως είπα και πριν, με αντίστροφη σειρά θα απαντήσω. Αν θα έπρεπε να υπάρχει μία μελέτη που θα κοιτάζει τη βιωσιμότητα και το δυναμικό που υπάρχει στην αγορά σε σχέση με τα best seller. Λοιπόν, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, τι είναι ακριβώς ο ηλεκτρονικός δανεισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα υποκατάστατο της πρόσβασης που έχει ένας αναγνώστης στα best seller. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο, μπορεί να πάει σε μια βιβλιοθήκη. Ε, πιστεύω πως ε, το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όσους δεν έχουν άλλη, άλλου είδους πρόσβαση. Επίσης μην ξεχνάμε πως οι βιβλιοθήκες έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό και δεν μπορούν ε, να ε, διαθέσουν κονδύλια, να αγοράσουν αρκετές ε, άδειε. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές το θέμα είναι να καλύψουν ένα καλό ποσοστό βιβλίων, ένα καλό ποσοστό πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένα βιβλία σε σχέση με κάποιο βιβλιοπωλείο, με κάποιο εμπορικό κατάστημα. Τώρα, τι θα κάνει η Επιτροπή για το ψηφιακό θεματολόγιο και για την πρόθεση του ηλεκτρονικού δανεισμού. Σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γνωρίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα από πολλές πτυχές. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, διότι υπάρχουν πιθανά ωφέλη αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ανάγκη πάντα να υπάρχει μία ε, λύση εκτός ε, νομικού πλαισίου, μία λύση πριν φτάσουμε στα δικαστήρια. Και πιστεύω πως χρειάζεται να εντοπίσουμε το πρόβλημα, δηλαδή να εντοπίσουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία κινούμαστε, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον και πώς μπορεί η συνεργασία μεταξύ εκδοτών και ε, βιβλιοθηκών να γίνει καλύτερη από ό,τι τώρα. Τώρα, ε, σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε για την πτώση του δανεισμού έντυπων βιβλίων στις κατοχώρες και με την αργία σταθερή αύξηση του ηλεκτρονικού δανεισμού. Πιστεύω πως η μείωση είναι περίπου 13 εκατομμύρια το χρόνο σε σχέση με αύξηση 1,3 εκατομμύρια ηλεκτρονικών βιβλίων. Ε, πιστεύω πως ε, καταρχάς να δούμε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό σε σχέση με τα έντυπα. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι ένα το κρατούμενο και επίσης υπάρχει και το θέμα του πόσο δημοφιλής είναι ο ηλεκτρονικός δανεισμός και ο δανεισμός έντυπων βιβλίων. Πώς αλλάζουν όλα αυτά. Και να πω επίσης και κάτι άλλο. Άκουσα τις ανησυχίες για τον ηλεκτρονικό δανεισμό και υπάρχει λοιπόν η ανησυχία ότι οι ε, δημόσιες βιβλιοθήκες προσφέρουν δωρεάν βιβλία σε σχέση με τα ηλεκτρονικά βιβλία που μπορεί κάποιος να αγοράσει. Δηλαδή κατηγορείται ότι διαταράσει την αγορά μια ε, βιβλιοθήκη. Εγώ θεωρώ πως είναι θέμα αναλογικότητας, δηλαδή αποδεχόμαστε τις ε, διταράξεις στην αγορά εργασίας ε, αλλάζοντας τις, ε, τα ημερομίσθια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως το σημαντικό είναι να αποφασίσουμε για τη σωστή ισορροπία, τη σωστή αναλογία, δηλαδή τι ποσοστό αναγνωστών μπορεί να καλύψει μία βιβλιοθήκη σε μία συγκεκριμένη κοινότητα, τι ποσοστό ε, υπάρχει διαθέσιμο σε ηλεκτρονικά βιβλία κτλ. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τις ανάγκες έτσι ώστε να μην υπάρχουν σοβαρές τρευλώσεις στην αγορά. Αλλά σίγουρα κάποιο ποσοστό είναι αναπόφευκτο. Αυτά. Νομίζω πως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Θα κάνω και εγώ κάποια συμπληρωματικά σχόλια. Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας σχετικά με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Να σας πω για τις κάτω χώρες, ο μεγαλύτερος διανομέας ηλεκτρονικών βιβλίων και σε βιβλιοπολία. και στο διαδίκτυο και στις ε, δημόσιες βιβλιοθήκες και στις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κανιβαλισμός ανάμεσα στο δανεισμό και στην πώληση βιβλίων. Κατά μέσο όρο δηλαδή, τα βιβλία που δανείζονται οι χρήστε μιας βιβλιοθήκη είναι βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από τρία χρόνια, ενώ τα βιβλία που πολλούνται είναι βιβλία που κυκλοφόρησαν ένα χρόνο πριν. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο θέμα, δεν κάνει βαλίζει μια χώρα την άλλη. Δεν ξέρω τι ε, γίνεται στις ε, άλλες χώρες, ε, αλλά νομίζω πως στη Δανία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, οι βιβλιοθήκες δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά τα πρόσφατα βιβλία, διότι οι διανομής δεν τους παρέχουν αυτά τα βιβλία. Στα ηλεκτρονικά βιβλία, μάλιστα, διατηρούν το δικαίωμα να μην τα διαθέτουν στις βιβλιοθήκες για κάποιο χρονικό διάστημα και υπάρχει μια παρόμοια ρύθμιση και για τα έντυπα βιβλία. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε. Και σχετικά με την ερώτηση, με την ερώτηση της κυρίας Φερχάιεν, να πω ότι καλό θα είναι να μην συγκρίνουμε με συγκεκριμένα νούμερα, διότι πράγματι έχει παρατηρηθεί μια πτώση στο δανεισμό έντυπων βιβλίων στις ε, δημόσιες βιβλιοθήκες τα τελευταία δέκα χρόνια στις κάτω χώρες. Όμως, μην ξεχνάτε και ότι στις κάτω χώρες υπάρχει μεγάλο ποσοστό δανεισμού ε, βιβλίων ανα, αναγνώστη σε σχέση με άλλες χώρες. Και ταυτόχρονα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, υπήρχαν και άλλες εξελίξεις, δηλαδή πειρατεία των ηλεκτρονικών βιβλίων, κάτι το οποίο άνθησε ε, το 2011 και 2012. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση στην πειρατεία ακριβώς επειδή υπάρχει νόμιμη προσφορά ηλεκτρονικών βιβλίων στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Στι κάτω χώρε πρέπει να πληρώσει για να γίνει μέλο σε μια βιβλιοθήκη. Μετά όμω μπορεί να δανειστεί όλου αυτού του 11.000 τίτλου που βρίσκονται στο σύστημα. Και έχουν γίνει και άλλε εξελίξει, όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι λίγο επικίνδυνο, θα έλεγα, να συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία. Χρειάζεται μια άλλη συζήτηση ε, που θα σταθεί και θα αφιερωθεί στι εξελίξει αυτέ, θα έλεγα. Τέλο, οι δημόσιε βιβλιοθήκε θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο για να δανείζουν βιβλία. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν σε μια δημόσια βιβλιοθήκη. Ας μην λοιπόν εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στο δανεισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Ε, σας ευχαριστώ καταρχάς για την παρουσία σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω εν συντομία να αναφερθώ σε κάποιες επίκαιρες και σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού, διότι η συζήτηση που γίνεται εδώ σχετίζεται και με την εκπαιδευτική, περιφερειακή πολιτική, πολιτική και έρευνα στον τομέα της ενίας αγοράς. Υπάρχει το πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό και μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων. Ο Φρανκ Χάισμανς συμπροεδρεύει εξάλλου ε, με ιδιαίτερα ε, ε, πρόσφορο τρόπο και επεξεργάζονται μεταξύ άλλων και το θέμα του ρόλου των δημοσίων βιβλιοθηκών, ε, κυρίως για τον ηλεκτρονικό δανεισμό σε 23 κράτη-μέλη και οι Νορβηγοί συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα υπρογνωμόνων και υπάρχουν 16, ε, πολύ, ε, ενδιαφέρουσες μελέτες που έχουν γίνει για διαφορετικά σενάρια και έχω και αντίτυπα φέρει μαζί μου, μπορείτε να ε, τα πάρετε αν θέλετε, αλλά και επιγραμμικά ε, στην, στον ιστότοπο Europa, στην βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμα επίσης. Υπάρχει διαφανώ διάλογο επίσης με την κοινωνία των πολιτών. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε το ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού για την ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων. Υπήρχε επίσης ε, συμμετοχή της βιβλιοθήκης ε, ε, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό με ικανοποίησε ιδιαίτερα και από το Δουβλίνο στην Ιρλανδία Βλέπουμε πολύ σημαντικό ρόλο της βιβλιοθήκης για την ενσωμάτωση των προσφύγων στις τοπικές κοινότητες. Βλέπουμε πόσο μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί η βιβλιοθήκη γιατί είναι ασφαλής τρίτος χώρος, ο δεύτερος χώρος όπου μπορεί κάποιος να αποκτήσει γνώσεις σχέση με τον πολιτισμό της χώρας σας. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. Φυσικά μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό το έγγραφο, αυτή τη μελέτη που μας είπατε. Ε, δεν ξέρω αν μιλώ και για τους άλλους συναδέλφους ε, ε όταν λέω πως ε, μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος αυτό το θέμα ε, κυρίως σε αυτό το τρίγωνο της ε, μετεκπαίδευσης ε, των ενηλίκων, ε, της παιδείας ε, στα μέσα και την πληροφορία, αλλά δεν ξεχνούμε φυσικά τη διάσταση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων θα μπορούσαμε ίσως και εμείς ως Επίτροποι να επιμβαθύνουμε σε αυτό. Ίσως ε, δεν το έχουμε συζητήσει. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και υπάρχει και πολύ υλικό προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες συστάσεις, ε, να δούμε κάποιες προπτικές. Έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συζητήσουμε και με αυτή την ε, ομάδα η οποία υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, αυτό το Reflection Group και να δούμε φυσικά και την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ε, θέματα τα οποία συζητούμε εμείς από καιρό. Για παράδειγμα, η φορολόγηση για τα ηλεκτρονικά βιβλία ε, και τι μπορεί να γίνει με τα βιβλία γενικότερα. Και υπάρχει και το γεγονός ότι ίσως στο παρελθόν να υπήρχε κάποιο πρόγραμμα το οποίο να ήταν ειδικά αφιερωμένο στις βιβλιοθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε προγράμματα τα οποία μπορεί να τις περιλαμβάνουν, αλλά δεν είναι συγκεκριμένη στόχευση σε αυτό. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι για την πολύ καλή συνεισφορά σας. Ε, έχουμε και ένα ε, σημείωμα. Ευχαριστούμε το Τμήμα Πολιτικής ε, για τα όσα έκανε και για το σημείωμα το οποίο μας ετοίμασε και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε κάτι θετικό. Τις προάλλες, στην πόλη μου, στη Ρώμη, πήγα ε, στα εγγένεια μιας βιβλιοθήκης μιας απομακρυσμένης περιφέρειας της Ρώμης εκεί για να γεννιάσω τη βιβλιοθήκη λοιπόν, ε, πρέπει να πω ότι ήταν μοναδική εμπειρία, διότι ήταν τεράστια η συμμετοχή του ε, ε, κόσμου σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, ενθουσιασμό, ενεργή συμμετοχή και ίσως να είναι και μεγαλύτερος από όσο θα είχαν δείξει αν είχαμε γενιάσει ένα εμπορικό κέντρο. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι μεγαλύτερος το κτίριο το πήραμε από την Καμόρα, από την οργανωμένη μαφία. Ε, κατασχέθηκε το κτίριο και αποφασίστηκε να το ε, μετατρέψουμε σε βιβλιοθήκη. Και το λέω αυτό διότι το θέμα των πόρων ε, του οργανωμένου εγκλήματος είναι πλέον και ευρωπαϊκά μέτρα. Δεν είναι οι μόνοι πόροι, αλλά θα μπορούσαμε και να το σκεφτούμε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε στην εθνική νομοθεσία, γιατί η εθνική νομοθεσία μας προβλέπει και κονδύλια για τις για τους Δήμους αλλά και για μη κυβερνητικούς κερδοσκοπικούς συγγνώμη, οργανισμούς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ολοκληρώθηκε αυτό το τμήμα της ε, συνεδρίασης. Ένα λεπτό για να περάσουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, αμέσως μετά έχουμε την έκθεση του συναδέλφου Κούρτσιο Μαλτέζα, αλλά ένα λεπτό μόνο για να αποχαιρετήσω τους καλεσμένους μας. Eh, Συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις εργασίες μας. Έχουμε τώρα το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Πρόγραμμα στήριξης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για το διάστημα 2017-2020. Εισηγητής είναι ο συνάδελφος Κούρτσο Μαλτέζε. Έχουμε σήμερα την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Ε, θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο αποφάσισε να εγκρίνει ένα κανονισμό για το πρόγραμμα στήριξης. Η χρηματοδότηση είναι περίπου 142 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια. Τα κράτη-μέλη βεβαίως μπορούν να αποφασίσουν να προσθέσουν και άλλη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα αυτό και η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα θέμα άλλωστε που αφορά τις περιφέρειες και μετά από ένα πρόβλημα που υπήρχε με την Επιτροπή ΕΚΟΝ, η ψηφοφορία με, ε, για την Επιτροπή ΡΕΤΖΙ είναι για, τις, για τα τέλη Νοεμβρίου. Εμείς ε, ζητήσαμε να έχουμε και γνωμοδότηση για του τομείς της εκπαίδευσης, ελπίζουμε και του πολιτισμού και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών Τετάρτη 29 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα. Να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Μάλτα για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς λοιπόν όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προέκυψε από κατόπιν προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για στήριξη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επί εθελοντικής βάσεως κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών και αναφερόμαστε σαφέστατα σε κάποιες εμπειρίες όπως την εμπειρία της Ελλάδας και της Κύπρου. Το αίτημα λοιπόν, είπαμε, είναι σε εθελοντική βάση από πλευράς κρατών μελών, αλλά αυτή στιγμής ενεργοποιηθεί αυτή η τεχνική στήριξη, η τεχνική στήριξη ε, υποδεικνύει ε, σε ποιους τομείς θα πρέπει να γίνει η παρέμβαση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ο πολιτισμός και η παιδεία. Και όλοι οι τομείς που αφορούν ε, την Επιτροπή μας δηλαδή. Η γνωμοδότησή μου, σεβόμενη και το θεσμικό ρόλο της Επιτροπής μας, είναι να ε, υπάρχει ε, μια εξαίρεση για την παιδεία και τον πολιτισμό όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Δηλαδή να επισημάνουμε την ιδιαιτερότητα των τομέων της παιδείας και του πολιτισμού που δεν ε, μπορούν να καλύπτονται από κριτήρια καθαρά οικονομικής απόδοσης, αλλά πρέπει να επιτυγχάνουν άλλους στόχους. Και ακόμα και όταν επιτυγχάνουν οικονομικής φύσεως στόχους, είναι πολύ πιο περίπλοκος και άμεσος, έμεσος με τον οποίο επιτυγχάνεται. Αυτό είναι η πρώτη μας ανησυχία. Δεύτερον, θέλουμε να αποφύγουμε η οικονομική πρικοδότηση αυτού του προγράμματος να προέρθει από πόρους οι οποίοι ούτως ή άλλως προορίζονται για την παιδεία και τον πολιτισμό. Και ξέρετε ότι ε, οι πόροι αυτοί δεν αρκούν ούτως ή άλλως, επομένως θα υπήρχε πρόβλημα εάν περιοριστούν περαιτέρω για να χρηματοδοτήσουμε άλλα πράγματα. Τρίτο θέμα, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τόσο κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ε, όσο και κυρίως για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, για να δούμε πώς λειτουργούν πιο συγκεκριμένα αυτά τα προγράμματα και να προσπαθήσουμε να έχουμε ενεργό συμμετοχή από πλευράς ε, κοινωνικών εταίρων, εγκαίρως, ώστε να μην διαπράξουμε σφάλματα τα οποία έχουν ε, υπάρξει στο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις εμπειρίες του παρελθόντος, ε, μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια συνέπεια στις της στα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ συχνά οι παρεμβάσεις στον τομέα της ε, παιδείας και του πολιτισμού ε, έχουν αποτελέσματα σε κάποιου τομεί. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει έχουν λειτουργήσει σε κάποιου τομεί, αλλά σε άλλου, όπω την παιδεία, έχουν δημιουργήσει πολύ επικίνδυνου περιορισμούς στην πρόσβαση στην παιδεία για διάφορα κοινωνικά στρώματα. Σε αυτά λοιπόν ε, ε αναφέρεται κυρίως η γνωμοδότηση. Ε, τα χρονοδιαγράμματα είναι αυτά τα οποία σας ανέφερε η Πρόεδρος και φυσικά ε, ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις και τις παρεμβάσεις σας ε, προκειμένου να μπορέσω και να πατήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Θέλει κανείς το λόγο. Ναι, ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να αναφέρω πόσο ε, ικανοποιημένος είμαι με αυτό το πρόγραμμα διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2020 Υπάρχουν αρκετά που έχουν ισχνή ανάπτυξη μετά την χρηματοπιστωτική κρίση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν έτσι ιδιαίτερο βάρος για την κοινωνική συνοχή, όχι μόνο για τα νομοθετικά ζητήματα. Ε, επιδοκιμάζω λοιπόν τις προτάσεις του εισηγητή. Θα ήθελα να σχολιάσω τα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, είναι ουδέτερα, ουδέτερη αυτή η πρόταση από δημοσιονομικής άποψης. Όμως θα πρέπει να μην δημιουργηθεί προηγούμενη για τη χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, η υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ετήσιας παρακολούθησης ε, για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του τρίτον. Ο στόχος είναι η απόκτηση ε, δεξιοτήτων και βοήθεια προς τους νέους, ώστε να έχουν κριτικό πνεύμα, να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τεχνική αρρωγή για ε, εκπαιδευτικά ζητήματα ή επιμορφωτικά ζητήματα. Και θα πρέπει να έχουν διακριτική ευκαιρία τα κράτη-μέλη να ζητούν αυτή τη βοήθεια. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοιχτό για ε, τα, τους φορείς ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Επικροτώ την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το άρθρο 5, διότι έτσι μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλα προβλήματα, όπως καταπολέμηση της στόχιας, προβλήματα που ανακύπτουν με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Ο κύριος Μαραγκάλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Μετά που άκουσα τόσα είπε ο κύριος Μαλτέζε, νομίζω ότι συμφωνώ και με τις ανησυχίες του και με αυτά τα οποία μας προτείνει στη γνωμοδότησή του. Θα ήθελα απλώς να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα το οποίο υφέρπει και σίγουρα θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ξεκινώντας από την εμπειρία των προηγούμενων ετών, ε, έχει γίνει ένα μάντρα. Η αυτόματη λύση, το ρητό, Κάθε φορά το χρησιμοποιούμε, το εφαρμόζουμε και θεωρούμε ότι είναι η πανάκια για όλα, αποδεδεγμένη αποτελεσματικότητα ε, και πάντα μπορεί να μας οδηγήσει στα κατάλληλα αποτελέσματα. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι πολιτικές αποδείχθηκαν ε, εντελώς αντιπαραγωγικές και εντελώς αντίθετες προς τους στόχους που θέλαμε να επιτύχουμε. Τα προγράμματα λοιπόν στήριξης ε, ξεκινούν από τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φαίνεται ότι υπάρχει ε, ε σχέση με την πολιτική συνοχή και τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης. Εάν τα ε, όλα αυτά μαζί, νομίζω ότι δεν θα πάμε σε σωστό δρόμο. Ο στόχος των πολιτικών συνοχής είναι και θα πρέπει να είναι η μείωση των ανισοτήτων. Τα μέτρα της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιορίσουν τις λεγόμενες ανισορροπίες, αυτό το imbalances που χρησιμοποιούμε συνέχεια στην ευρωπαϊκή ορολογία. Το να μην ε, χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα μέτρα για τους δύο στόχους δεν είναι μόνο επικίνδυνο, αλλά είναι και ρηψοκίνδυνο και από κοινωνική σκοπιά αλλά και ε, όσον αφορά τις πολιτικές που υποτίθεται ότι προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Συνοχής. Συμφωνώ με τον κύριο Μαλτέζε και τις ανησυχίες που εξέφρασε όσον αφορά τις πολιτικές παιδείας, πολιτισμού και το καθεξής και θα πήγαινα και ένα ε, βήμα παραπάνω. Εάν τις εξετάζουμε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι κάνουν οι χώρες μέλη για να προωθήσουν την παιδεία, για να προσθέσουν ε, τι ε, λαμβάνουν υπόψη τους όσον αφορά την πολιτική συνοχή σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, κατάρτισης και το καθεξής και πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερη σημασία σε αυτές τις πολιτικές. Και επίσης ποια κονδύλια της συνοχής ε, ε, μπορούμε να τα αφιερώσουμε σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι λίγο ύποπτη η σύμπτωση ε, που υπάρχει στα θέματα αυτά με την εμφάνιση μηνυμάτων που αυξάνεται συνεχώς, που αναφέρονται σε αλλαγή στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, κάνουμε τμήμα της χρηματοδότησης χρηματοδοτικά μέσα. Χρηματοδοτικά μέσα τα οποία υποτίθεται ότι είναι το σχέδιο Juncker και λοχεύει ο ίδιος κίνδυνος εδώ. Να συγχύσουμε τους στόχους και τις πολιτικές που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναφερόμαστε και σε κριτήρια γιατί να μην περάσουμε από τα κριτήρια που αφορούν κυρώσει σε όσοι δεν συμπεριφέρονται καλά, στα κριτήρια που ενισχύουν ε, με βάση επενδύσεις και με βάση ε, δυνατότητες της κάθε χώρας. Ε, που νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όταν προσπαθούμε να μειώσουμε τις ανισότητες. Νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε σε αυτό και εδώ νομίζω ε, ε, θα υποβάλουμε και εμείς κάποιες τροπολογίες οι οποίες πιστεύω ότι συνάδουν με αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Μαλτέζε και ελπίζω να μπορέσουμε και εμείς με τη γνωμοδότησή μας ως Επιτροπή Προελδισμού να συνεισφέρουμε στην έκθεση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή ο Λουίτζι Μόργανο. Νομίζω ότι ο συνάδελφο Νέκοφ ε, ήδη ω και ο εξέφρασε την άποψη τη ομάδα μα. Νομίζω ότι Πρέπει να σας πω ότι εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες ε, που εκφράστηκαν από τον Κούρτσιο Μαλτέζε, ιδίως ε, το δικαίωμα στην παιδεία, η στόχοι της παιδείας και της κατάρτισης και αν καταφέρουμε με βάση της τροπολογίας να επενθυμίσουμε αυτή την έννοια, η οποία πολλές φορές όταν ε, τη συζητούν κάποιες ε, ε, επιτροπές επί του θέματος θα το αναφέρουν ως δαπάνη και όχι ως επένδυση. Και νομίζω ότι κάτι θα μπορούσαμε να έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να μειώσουμε περαιτέρω λοιπόν ε, μια παρέμβαση που ούτω ή άλλω είναι ήδη περιορισμένη και νομίζω ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο αν μας περιορίσουν και άλλο του πόρους. Εάν λοιπόν αποκλείσουμε τα κονδύλια αυτά από τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων νομίζω ότι ε, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών διότι η ε, η συζήτηση αυτή θα αφορά απλώς και μόνον ε, ένα μερικό τμήμα ε, και θα είναι μόνο μια πολύ περιορισμένη ανάγνωση. Και νομίζω ότι αυτό το εκφράζουμε και με την τροπολογία παριθμών 10. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Θα... Ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση στο συντάκτη, αλλά η κυρία Αντινόλφη πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μαλτέζε για την γνωμοδότηση. είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το επαναλαμβάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την παιδεία ως αμελιώδης δικαίωμα. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντε συνάδελφοι, όπως επίσης συμφωνώ με το συνάδελφο Μαλτέζε ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την εξήγηση που εξηγεί πώς τα προγράμματα προσαρμογής τα οποία εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες φορές μείωσαν ε, τη δαπάνη στον τομέα της παιδείας και της κατάρτισης. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Συμφωνώ ότι δεν πρόκειται για δαπάνη αλλά είναι επένδυση ε, και για άλλη μια φορά όμως ε, διαπιστώνουμε ότι το χρηματοδοτικό σκέλος, αν μου επιτρέπετε, ε, αντιμετωπίζει πολύ μειοπικά τα θέματα όταν αφορά θέματα παιδείας και εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ναι, δεν τα καταφέρνουμε να περάσουμε την άποψή μας, αλλά αυτά τα προγράμματα, αυτή η χρηματοδότηση, τα μέτρα τα οποία εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησαν σε μια πάρα πολύ αυστηρή λιτότητα σε κάποιες χώρες και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπήρξαν φρικτά αποτελέσματα μετά από τα χρόνια μέτρων λιτότητας και Οι ζημιωμένοι φυσικά ήταν ε, ε, οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τα παιδιά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ανακάμψουν και ποτέ. Ελπίζω λοιπόν ότι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε θα είναι προς το γεγονό ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα που, τα οποία πρέπει να ε, προστατεύσει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην παιδεία, αλλά υπάρχουν και θέματα όπως η υγεία των παιδιών, τα οποία δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε. Ελπίζω να συνεργαστώ και εγώ με τους υπόλοιπου συναδέλφου και ευχαριστώ και πάλι τον ε, συντάκτη τη γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου. Αν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, θα ήθελα και εγώ να πω την άποψή μου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν όντω το ερμηνεύουμε έτσι, ότι αποκλείονται η παιδεία και ο πολιτισμός και αν όντω ε, προέβλεπαν τα κονδύλια και την συμπερίληψη, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ με την κυρία Τινόλφη, είναι επενδύσει αυτά τα πράγματα και σε άλλες περιπτώσεις ε, ε, θέλαμε να μην προσμετρηθούν από τον υπολογισμό στον προπολογισμό, τα κονδύλια για την παιδεία και την πολιτιστική καινοτομία. να μην θεωρούνται λοιπόν ε, ε, τμήμα των τακτικών δαπανών. Ε, και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η τροπολογία η οποία αναφέρεται στην πρόσβαση στον πολιτισμό. Πρόσβαση στην παιδεία λοιπόν και πρόσβαση στον πολιτισμό. Θα ήθελα να καταλάβω το εξή. Επειδή προηγουμένω ο κύριος Μαραγκάλ είπε ότι θα μπορούσαμε ίσω να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω. Αυτή είναι ερώτηση. Εγώ δεν κατάφερα να το εξετάσω περαιτέρω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προωθήσουν αυτές τις ε, ε, πλατφόρμες ε, για την εκπαίδευση, για την τον πολιτισμό, τη ε, δημιουργική βιομηχανία, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μεν εξετάζεται, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ αμφίσιμα τα πράγματα και ασαφή. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε κάποιες επενδύσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είναι αφιερωμένες στο τομέα αυτό, για να υποστηρίξουν αυτούς τους τομείς, οι οποίοι είναι παραμελημένοι. Δηλαδή, όχι μόνο να μην υπάρξουν περίπτωκοπές, αλλά να ζητήσουμε κιόλας ε, να συμπεριληφθούν. Είμαστε στη διαδικασία των τροπολογιών. Μια πρόταση ήθελα να κάνω. Αν συμφωνεί και ο συντάκτης, ίσως θα μπορούσαμε να το ε, διευκρινίσουμε λίγο ακόμα αυτό. Ναι, ο κύριος Μαλτέζε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική αυτή η πρόταση. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι νομίζω ότι είχαμε μια συζήτηση, ε, κοινή συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί διχασμούς. Το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, κατά την άποψή μου, περιβάλλεται και από υπερβολικές ρητορίες και ιδεολογίες. Εγώ προσπάθησα να σταθώ στα πιο ρεαλιστικά στοιχεία, διότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ένα τεχνικό εργαλείο στη διάθεση των κρατών μελών στην πραγματικότητα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πού έχουν αποτελέσματα και πού δεν έχουν αποτελέσματα. Η εμπειρία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μας δείχνει ότι στις χώρες της Νότιας Ευρώπης τις οποίες εφαρμόστηκαν και όπως αναφέρονται και στο έγγραφο, ιδίω ε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι παρεμβάσεις στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού ήταν παρεμβάσεις οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα διότι ουσιαστικά απλώς έγιναν περικοπές. το να γίνονται περικοπές και να γίνεται μια διαδικασία εξέτασης των δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να είναι και ενδιαφέρον, διότι μπορεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πούν πού μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις όταν δεν είναι παραγωγικές και καρποφόρες οι δαπάνες σε δημόσιο επίπεδο. Αλλά το να το βασίσουμε μόνο σε αυτά τα θέματα είναι ε, επικίνδυνο, επιζήμιο, αλλά είναι λανθασμένο και ως αρχή, γιατί η παιδεία είναι δικαίωμα και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Είναι λανθασμένο όμως και σε οικονομικό επίπεδο, διότι σε χώρες όπως την Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω και την Ιταλία, την Ισπανία, χώρες ε, στις οποίες ε, τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και του δημοσίου χρέους έγιναν μεγάλες περικοπές στην παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε ένα μέσο επενδύσεων, όπως έλεγε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι στις χώρες της Νέτιος Ευρώπης ανακόπτουμε την ε, κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή είναι από τα βασικά μέσα δημιουργίας πλούτου, παραγωγής, ε, δημιουργικότητας, ευημερίας και αυτό τελικά συνέβη. Και πρέπει να ε, καταγράψουμε πώς λειτουργήσαν αυτές οι πολιτικές και να μην το έχουμε ως λάβαρο για να υποστηρίξουμε την τάδη τη δυναθέση. Θα πρέπει λοιπόν στην παιδεία να παρέμβουμε με άλλα κριτήρια. Θα πρέπει να καθορίσουμε άλλες γραμμές παρέμβασης. Και επίσης όσον αφορά την οικονομική χρηματοδότηση νομίζω ότι όλοι ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα ήταν αντί τροφά, πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε, να αυξήσουμε τους πόρους και όχι να τους περικόψουμε κι άλλο και να τους χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι, το είπα και προηγουμένως, 29 έκτου, 5 και μισή το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαλτέζε και να περάσουμε Συγγνώμη, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να σα πούμε ότι αύριο θα συνεχίσουμε στις 9 ακριβώς. Με πλούσια ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε ε, τώρα με τη συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών και επειδή έχουμε και λίγη ώρα στη διάθεσή μας, ε, η πρόεδρο. αύριο θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας και πέντε λεπτάκια διάλειμμα ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν και όσοι δεν θα παραμείνουν και θα ήθελα να παραμείνουν μόνο οι συντονιστές και όσοι ε, άλλοι επιτρέπεται να συμμετέχουν. Ευχαριστώ.